Colleagues, um, we were... Συνάδελφοι, περιμέναμε έναν ακόμα από τους συμμετέχοντες και μια ανακοινώση που θα τη λάβετε και σε email όλοι στα γραφεία σας. Η παγιματινή συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις, στις 3 και μισή και όχι στις 3. Το επαναλαμβάνω, η απογευματινή συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 3.30 και όχι στις 3. Το email θα πάει σε όλα τα, τα γραφεία όλων σας και επίσης η ψηφοφορία αναβάλλεται ως την επόμενη Δευτέρα. Την επόμενη ε, Δευτέρα στις 5.30 και πάλι θα ενημερωθείτε και με email. Παρακαλώ λοιπόν ενημερώστε τους συναδέλφους σας ότι η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 3 αλλά στις 3.30. Να έρθουν λοιπόν τις ψηφοφορίες στις 3.30. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να οργανωθείτε καλύτερα. Γιατί είναι αρκετοί εκείνοι που δεν μπορούσαν να είναι εδώ στις 3. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για να οργανωθούμε έτσι και να αναβάλουμε την ε, άλλη ψηφοφορία ως τη Δευτέρα. Στείλαμε mail λοιπόν σε όλους, αλλά φροντίστε και να ενημερώσετε τους πάντες. Είναι όλοι οι συμμετέχοντες εδώ. Ωραία, ας ξεκινήσουμε. Με συγχωρείτε συνάδελφοι για την καθυστέρηση, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Αυτή τη σημαντική ακρόαση, έρευνα για την εικαζόμενη μεταφορά και παράνομη κράτηση προσώπων από την CIA. Έχουμε συμμετοχή της κυρίας Ραλούκα Ραντέσκου από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σπουδών, Πολιτικών Σπουδών, την ε, συναδελφά Βαζολή από την Επιτροπή τη δική μας, τον κύριο Κρόφτον Μπλακ από τον Οργανισμό Ερευνητικής Δημοσιογραφίας και εδώ θα δούμε το πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό της έρευνας για το τι συνέβη με τις εικασίες, με τις εικασίες μεταφοράς και παράνομης κράτησης ε, φυλακισμένων σε ευρωπαϊκές χώρες από την CIA. Το πρόβλημα έχει οδηγήσει σε επανειλημμένες καταγγελίες αυτής της μυστικής κράτησης και έκτακτης παράδοσης και του συνολικού προγράμματος με πολλαπλές παραβιάσεις ανθρωπινών δικαιωμάτων. Ε, μιλάμε για τα ψηφίσματά μας 14 Φεβρουαρίου 2007, 11 Σεπτεμβρίου 2012, 10 Οκτωβρίου 2013 και 11 Φεβρουαρίου 2015. Θα θυμάστε αυτή τη σημαντική έρευνα για τις παραδόσεις ε, της CIA. Ε, ο κύριος Κοέλιου ήταν υπεύθυνο. Σήμερα έχουμε τη συνέχεια αυτής της σημαντικής έρευνας που παρακολουθούν οι συντονιστές μας. Δεν θέλω να καθυστερήσω κι άλλο, αλλά να περάσουμε απευθείας στις παρεμβάσεις των ε, συμμετεχόντων. Να ξεκινήσει λοιπόν αυτή η πρωινή συζήτηση για να ενημερωθούμε στην Επιτροπή μας για το που έχει φτάσει αυτή η σημαντική έρευνα και από την Αμερικανική πλευρά αλλά πάνω απ' όλα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκινούμε λοιπόν την πρωινή συνεδρίαση με την παρουσίαση του εγγράφου που αφορά την έρευνα από την κυρία Έλσπεθ Γκάιλτ και την Αλούκα Ραντέσκου από το ΣΕΠΣ το Κέντρο για τις Ευρωπαϊκές Σπουδές Πολιτικής. Έχετε το λόγο, κυρίες μου. Ευχαριστώ πολύ τον Πρόεδρο της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Ευχαριστώ την Επιτροπή στο σύνολό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γνωρίζουμε καλά την σημασία των εργασιών της Επιτροπής σας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην αναζήτηση απαντήσεων στις ερωτήσεις που έχουν τεθεί με την τραγική παραβίαση του κράτους δικαίου όσον αφορά τις δραστηριότητες ε, καταπολέμησης της τρομοκρατίας που έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ άλλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το διάστημα 2002 έως 2007. Μας ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσουμε τι έγινε όσον αφορά την λογοδοσία και να εξετάσουμε τι έχει γίνει όσον αφορά την συνενοχή κρατικών φορέων σε έναν αριθμό κρατών μελών στο ε, πρόγραμμα ε, έκτακτης παράδοσης ε, και μυστικής κράτησης της CIA, το οποίο έχει επικρίνει και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και άλλοι σημαντικοί παράγοντες στην κυβέρνηση και τη γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει γίνει σημαντική έρευνα των παράνομων δραστηριοτήτων της CIA ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, μεταφορά ανθρώπων ε, και την κράτηση ανθρώπων. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μάλιστα μίλησε για βασανισμό. Εξετάσαμε ποια ήταν η αντίδραση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις έρευνες που έχουν να κάνουν με αυτές τις παράνομες δραστηριότητες και που ε, αντίκυνται στις ε, διεθνείς δεσμεύσεις μας και στο διεθνές δίκαιο. Θα γνωρίζετε φυσικά ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν συνυπογράψει τη Σύμβαση των Ηνωμένων ε, Εθνών για... κατά του βασανισμού. Ε, δεσμεύονται λοιπόν να ερευνήσουν οποιασδήποτε κατηγορίες ε, για βασανισμούς. Θα πρέπει όμως να ερευνούν και οποιασδήποτε άλλες δραστηριότητες όταν υπάρχει κάποια υποψία ότι άτομα εντός ε, της δικαιοδοσίας μας ε, συμμετείχαν σε τέτοιες δραστηριότητες. Έχουμε λοιπόν πολύ ισχυρή υποχρέωση που έχει την νομική βάση στο διεθνές δίκαιο Έχουμε επίσης υποχρέωση να παράσουμε όσο γίνεται αποκατάσταση στα ε, θύματα. Τι έχει γίνει λοιπόν. Τα δύο πιο πρόσφατα στοιχεία που έχουν ανακύψει μέσα στο τελευταίο δεκάμινο είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Το πρώτο στοιχείο είναι δύο αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πρόκειται για τις αποφάσεις Αλνασίρη και Αμπού Ζαμπάιντα ε, του Ιουλίου του 2014 και οι δύο αφορούσαν την Πολωνία. Οι αποφάσεις ε, ήταν ιδιαίτερα μακροσκελής, 150 ε, σελίδες και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων ε, Δικαιωμάτων ε, αναφέρεται στον βασανισμό των ε, ανθρώπων αυτών με την συνενοχή της πολωνικής κυβέρνησης που επέτρεπε στην CIA να έχει κέντρο μυστικής κράτησης στο έδαφος της. Το δικαστήριο διαπιστώνει ποια είναι τα γεγονότα και επίσης ότι η κυβέρνηση της Πολωνίας ε, δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της. Τίθεται και το θέμα του άρθρου 13, αλλά η απόφαση αυτή δείχνει πόσο απαραίτητη είναι μια έρευνα καθώς και η δίωξη των υπευθύνων. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο που καλύπτουμε στην έκθεσή μας είναι η μελέτη της ε, Επιτροπής Πληροφοριών της ε, Γερουσίας ε, των Ηνωμένων Πολιτειών που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2014 και που με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες περιγράφει την έκταση των δραστηριοτήτων της CIA όσον αφορά βασανισμούς βασανιστήρια. Μας δίνει όμως και μια εικόνα όσον αφορά τη συνενοχή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στις ε, συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Η CIA επέλεξε να βασίζεται σε Ευρωπαίους συναδέλφους αντί για ε, στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε όλο τον κόσμο Και γιατί η CIA το επέλεξε αυτό. Διότι ακόμα και κατά την έναρξη του προγράμματος, ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών είχε σημαντικές αμφιβολίες όσον αφορά την νομιμότητα του προγράμματος αυτού. Θα δώσω τώρα το λόγο ε, στην συνάδελφό μου για να σας μιλήσει για το θέμα της λογοδοσίας. Ευχαριστώ πολύ. Να πω πώς θα προχωρήσουμε μελετήσαμε τις πληροφορίες μετά την κοινοβουλευτική μελέτη της κυρία Φλότ και είδαμε το κατά πόσο υπάρχει συνενοχή κάποιων κατών μελών στο πρόγραμμα παραδόσεων της CIA και από το φως των νέων εξελίξεων όπως το γεγονός ότι έκτοτε τουλάχιστον τέσσερα, τέσσερις παρανομές κρατήσεις επιβεβαιώθηκαν δύο στη Λιθουανία, μία στην Πολωνία και μία και μία στη Ρουμανία. Ε, κάναμε έρευνες για να δούμε αυτοί οι παράνομοι τόποι κατά πόσον ε, υπάρχουν εκεί. Επίσης στην Φύρομ βρήκαμε ε, κάποια στοιχεία και στοιχεία για την Λιθουανία, Ιταλία και Ρουμανία. Υπάρχουν διαφορετικοί λοιπόν βαθμοί συνενοχή των κρατών μελών στο παράνομο πρόγραμμα αυτό της CIA, είτε με ενεργό συμμετοχή, είτε με παθητική στάση και ανοχή. Σε κάποιες περιπτώσεις λοιπόν επέτρεψαν τις εσωτερικές πτήσεις στον εθνικό τους εναέριο χώρο κάποιες χώρες. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ως προς αυτό συνεργάστηκαν είτε παρήχαν πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες για την παράδοση των ε, προσώπων που μεταφέρονταν. για την περίπτωση που υπήρχαν υποψίε τρομοκρατική ενέργεια στην περίπτωση τη Ιταλία, λόγω χάρη το Ηνωμένο Βασίλειο. Βέβαια σε κάποιε χώρε εντοπίστηκαν τόποι παράνομη κράτηση, όπω αυτή που ανέφερα στη Λιθουανία, την Ρουμανία και την Πολωνία. Τα επίσημα έγγραφα που τα εξέτασε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιβεβαίωσαν τα γεγονότα. Και έτσι κοιτάξαμε την λογοδοσία. Μπορείτε να κοιτάξετε, να περάσετε στην, την προηγούμενη διαφάνεια. Εξετάσαμε τη λογοδοσία σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. Ως προς την εθνική διάσταση, είδαμε τις πολιτικές ε, έρευνες, τις δικαστικές έρευνες, τις ανακρίσεις, Και υπήρξε και μελέτη από το 2012 από το δικό μας κέντρο προς το Κοινοβούλιο όπου είδαμε και τις... Δεν είδαμε, δεν, υπήρξαν, δεν είδαμε στοιχεία από τον διαμεσολαβητή γιατί δεν υπήρξαν τέτοια. Απλώς το πώς εξετάστηκαν υποθέσεις στο δικαστήριο των ανθρωπινών δικαιωμάτων με την εμπλοκή της Πολωνίας. Επόμενη διαφάνεια, έτσι κατάσταση Ω προ τι εθνικέ και υπερεθνικέ έρευνε, στα πέντε κρατημέλη που επιλέξαμε ω πιο ενδιαφέροντα για τη μελέτη, όπως βλέπετε τέσσερις από τις εμπλεκόμενες χώρες ενεπλέξαν σε υποθέσεις που εξετάστηκαν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο οι εθνικές έρευνες σε δικαστικό ή πολιτικό επίπεδο βρίσκονται σε εξέλιξη και η εικόνα είναι αρκετά ετερογενής σε ό,τι αφορά το βαθμό συνενοχής και την πραγματική λογοδοσία. Και στα πέντε κράτη-μέλη που ανέφερα και που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα αυτή, η έρευνα σε πολιτικό επίπεδο σε επίπεδο γενοβουλευτικό ή εκτελεστικό έχουν ολοκληρωθεί και οι κυβερνήσεις, τα κοινοβουλευτικά σώματα σε μεγάλο βαθμό έχουν αρνηθεί τη συμμετοχή του σε αυτό το πρόγραμμα παραδόσεων. Παρόλο που υπάρχουν αποδεκτικά στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν το αντίθετο. Οι δικαστικές ανακρίσεις έχουν διεξαχθεί και στα πέντε κράτη-μέλη που ανέφερα Και για να σας δώσω μια εικόνα κατά προσέγγιση του πώς έχουν τα πράγματα, έχουμε εντοπίσει έρευνες σε πολιτικό επίπεδο και στα πέντε κράτη-μέλη. Όμως ο πραγματικός χαρακτήρας και το πεδίο της κάθε διαδικασίας έρευνας ενδιαφέρει από τη μια χώρα στην άλλη. Σε δύο από τις πέντε χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία, είτε σε κυβερνητικό είτε σε κυβερνητικό επίπεδο έχουν υπάρξει έρευνες. Οι δικαστικές ανακρίσεις έχουν ολοκληρωθεί σε εθνικό επίπεδο, αλλά καμία δεν είχε κάποιο πραγματικό αποτέλεσμα. Λόγω χάρη στην Πολωνία, τον Ρωμανό Βασίλειο, την Ιταλία και τη Λιθουανία, η ποινική έρευνα εκκρεμεί ως προς την εκδικασία της εκτός από την Ιταλία. και οι αστικές προσφυγές έχουν υποβληθεί στην Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Να επικεντρωθώ... Να επικεντρωθώ στο γεγονός ότι οι έρευνες αυτές έχουν μεγάλου φραγμού ω προ τη λογοδοσία και αν ε, αναφερθούμε στα πρότυπα κάποιου δικαίου που έχουν προκύψει από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ιδίω λόγω τη υπόθεση τη Πολωνία, φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι καμία πραγματική έρευνα ουσιαστικά δεν έχει λάβει χώρα σε κανένα από τα κράτη-μέλη που αναφέραμε. Το πρόβλημα με τις έρευνες αυτές είναι διτό. Πρώτα απ' όλα, η απουσία, η έλλειψη ανεξαρτησίας των φορέων που εμπλέκονται στην έρευνα και το γεγονός ότι πολλά από τα κράτη-μέλη έχουν επικληθεί το δόγμα του κρατικού απορρίτου για να αποφύγουν την εργοδοσία και να αποφύγουν επίσης το να παραδώσουν τις απαραίτητες αποδείξεις για να ολοκληρωθεί σωστά η έρευνα. Στην επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Έχουμε λοιπόν νέα αποδεκτικά στοιχεία ότι υπάρχουν σοβαρέ ελλείψει στο κράτο δικαίου και στι ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούσαμε τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι θα υπάρξει ασυλία για τους Αμερικανούς που έχουν εμπλακεί στα βασανιστήρια των ε, φυλακιζόμενων, των κρατουμένων στα πλαίσια του προγράμματος αυτού. Δεν έχουμε ανάλογες δηλώσεις βεβαίως από Ευρωπαίους πολιτικούς ηθήνοντες, διότι αυτό θα ήταν αντίθετο με τις υποχρέσεις που έχουμε να αναλάβει λόγω της ε, Ευρωπαϊκής Σύμβασης, της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά των βασανιστήριων και του όλου καθεστώτος που επικρατεί για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε βασανιστήρια να έχουν όντως διεξαχθεί από τις Αμερικανικές Αρχές και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μας έχει δείξει τι βαθμό συνενοχής υπήρξε από κάποιους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως των υπηρεσιών τους. Και η Ραλούκα σας έδειξε συνολικά το πρόβλημα της περιορισμένης, της δειλής αντίδρασης των κρατών μελών στο να διεξάγουν πραγματικές έρευνε Αυτό είναι κατανοητό σε έναν βαθμό, διότι κάποια κράτη-μέλη θεωρούν ότι απλώς βοηθούσαν τους Αμερικανούς και ότι δεν είναι λάθος μας. Αυτή ήταν η αντίδρασή τους το 2003 και 2005. Οι Σουηδικές αρχές εντόψαν την πρώτη υπόθεση, η οποία έφτασε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την Επιτροπή του ΙΕ κατά των Βασινιστήριων. Παρ' όλα αυτά, η συνενοχή είναι ένα σημαντικό μέρος της όλης διαδικασίας. Όπως ανέφερα προηγουμένως, η έκθεση Feinstein καθορίζει πως και άλλοι Αμερικανοί φορείς, όπως ο Αμερικανικός στρατός, δίστασαν και τελικώς δεν ενεπλέξαν. Αν οι Ευρωπαϊκοί ε, οι Ευρωπαίοι είχαν αποφύγει να, να εμπλακούν, όπως συνέβη σε κάποια κράτη-μέλη, ίσως αυτές οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να μην είχαν λάβει χώρα. Επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Ραλούκα, θες να πεις τίποτα για το άρθρο 38? Ναι, ως προς την λογοδοσία και τις σχετικές απαιτήσει εντοπίσαμε τα πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως έχουν αναπτυχθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το πλαίσιο γιατί είναι η πρώτη φορά που κάποιο δικαστήριο βρίσκει την Πολωνία να έχει παραβιάσει τις αρχές του άρθρου 38 λόγω μη συμμόρφωσης από την πλευρά της πολωνικής κυβέρνησης με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτό και από τη σύμβαση. Η διάταξη αυτή απαιτεί οποιοδήποτε κράτος το οποίο έχει συμβληθεί στην χάρτα να παρέχει τις απαραίτητες διευκολύνσεις και τα απαραίτητα αποδεκτικά στοιχεία για την διερεύνηση μιας εκκρεμούσας υπόθεσης. Αυτό δεν συνέβη στις περιπτώσεις των ε, δικών των αγωγών κατά της Πολωνίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και είναι πρώτη φορά που θεώρησε το δικαστήριο ότι ένα κατεσμένος ε, έχει παραβιάσει το άρθρο 38. Εάν δει κανείς την απόφαση λεπτομερώς, βλέπει ότι υπάρχει ε, ένα, μια, ένα σύνολο από πρότυπα για το κράτος δικαίου και πώς πρέπει να διεξάγεται μια έρευνα. Θα πρέπει να είναι αυτή επίσημη, ε, ταχεία και ε, διεξοδική θα πρέπει να μην εξαρτάται από την εκτελεστική εξουσία, να περιορίζεται ή να αποφεύγει τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας ή το κυβερνητικό δόγμα του κρατικού απορρίτου, δηλαδή ουσιαστικά μια έρευνα θα έπρεπε, εάν το κράτος μέλος επικληθεί αυτό το δόγμα, επικαλεστεί μάλλον αυτό το δόγμα, να ε, μην υπάρχει άρνηση πρόσβασης στις πληροφορίες παρόλα αυτά. Αυτό το θεωρούσαμε πολύ σημαντικό εν ώψη των εμποδίων προς τη λογοδοσία που έχουμε εντοπίσει στα πέντε κράτη-μέλη που εξετάσαμε. Επόμενη διαφάνεια. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα. Το πρώτο, εμείς πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ηγηθεί ε, σε ε, ένα αίτημα να τοποθετηθούν επίσημα τα κράτη-μέλη για να ε, δούμε ποια είναι τα εμπόδια για τη λογοδοσία και για την δικαιοσύνη για τα θύματα, να ζητήσει να γίνει μια επίσημη έρευνα για να διαπιστωθούν οι ευθύνες. Δεύτερον, τακτικός διαρθρωμένος διάλογος χρειάζεται με τους ομολόγους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό θα ήταν μια εξαιρετική ιδέα για να δεσμεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταλλάσσει πληροφορίες. Η ανταλλαγή πληροφοριών που έγινε ε, μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών ε, των Ηνωμένων Πολιτείων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέκαμψε πλήρως στους δημοκρατικούς θεσμούς ε, και στις δύο πλευρές. Ε, ε, χρειάζεται οπωσδήποτε έλεγχος από θεσμικά όργανα ε, των ζητημάτων αυτών. Και ένας επαγγελματικός κώδικας δεοντολογίας για το χειρισμό τέτοιων στοιχείων και δεδομένων, ορίζοντας σαφώς τα κρατικά μυστικά και την κρατική ασφάλεια. Αυτό το έχουμε υποβάλει και γραπτός. Είδαμε την περασμένη εβδομάδα την απόφαση του δικαστηρίου στην υπόθεση ΣΡΕΜΣ. Ε, για θέμα ε, προσωπικών δεδομένων και πόσο παραβιάζεται ε, το κράτος δικαίου. Αυτά τα πράγματα, βασανιστήρια και έκτακτες παραδόσεις είναι παράδεκτα. Σε τακτά χρονικά διαστήματα επίσης θα πρέπει να αξιολογείται η συμμόρφωση των κρατών μελών με τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου υπό το νέο μηχανισμό της Κοπενχάγης και το νέο κύκλο πολιτικής. Ε, ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να επαγρυπνούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κάνουμε ακριβώς γιατί έχουμε τέτοιες προβληματικές καταστάσεις. Τελευταία σύστασή μας για τη λογοδοσία είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει αποτελεσματική και ουσιαστική δικαστική έρευνα ε, στο πόρισμα της έκθεσης Feinstein που λέει ότι η CIA πλήρωσε ε, πολύ υψηλά ποσά, πολλές φορές ε, δεκάδες εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών και μάλιστα μετρητά στις μυστικές υπηρεσίες και αρχές των, μελών, των κρατών μελών που ενέχονται και ε, αυτά αντιστοιχούν και σε ισχυρισμούς διαφθοράς. Είναι πολλά τα ποσά, πολύ μεγάλα τα ποσά που άλλαξαν χέρια, ε, μετρητά και σε αεροδρόμιο κοντά στη παράνομη φυλακή. Με διάφορες δικαιολογίες, χωρίς λογοδοσία, χωρίς αποδείξεις, μαύρα και παράνομα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you very much, uh, Professor Ευχαριστώ πολύ καθηγητά Κάλτ και δόκτωρ Ραντέσκο. Μας παρουσιάσατε ε, τη θέση των κρατών ε, μέλων. Στην αρχή, ίσως έπρεπε να πω ότι το Δεκέμβριο ε, του 2014 εκδόθηκε ε, αυτή η έκθεση στις ΗΠΑ που οδήγησε στη σημερινή μας ακρόαση. Το λέω αυτό για να ακούνε όσοι είναι εκτός της αίθουσας ε, το πλαίσιο και να γνωρίζουν που βρισκόμαστε. Πάμε τώρα στο επόμενο τμήμα της προάσης. Θα ακούσουμε την κυρία Εύα Ζολή που είναι μέλος της Επιτροπής ΛΥΒΕ και ήταν και μέλος της αντιπροσωπείας που μετέβη στο Βουκουρέστι πριν από λίγες εβδομάδες και ε, εξέτασε τους ισχυρισμούς για και τις κατηγορίες για τη Ρουμανία και θα μας εξηγήσει το επόμενο τέταρτο τα ευρήματα και τα απορίσματα της Επιτροπής εκεί. Ε, της Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους σας. Πρέπει να πω ότι συμμετείχα σε αυτή την αντιπροσωπεία, σε αυτή την αποστολή, μαζί με την Τάνια Φαγιόν, τη Λόρα Φεντέρα, το Γιουρούν Λέναρτς και την κυρία Ραμόνα Νικόλ Μανέσκου ε, που είναι μέλος ε, από τη Ρουμανία και μας συνόδευε. Στην αρχή ήμουν πολύ αισιόδοξη ότι με την έκθεση αυτή της γερουσίας, ακόμα και αν δεν κατονομάζονται χώρες, αν έχουν διαγραφεί τα ονόματα, ξέρουμε ότι έχει κάνει δουλειά και η Διεθνής Διαφάνεια και όμιλο Όμιλος Δημοσιογράφων της Ερευνητικής Δημοσιογραφίας κατάφεραν να ανακτήσουν τα ονόματα των χωρών και ήταν και εύκολο να βρούμε σε τι αντιστοιχούσε ε, η μαύρη κοιλίδα, το όνομα που είχε διαγραφεί στην έκθεση Φάινστάιν ήταν η Ρουμανία. Και θεωρούσαμε ότι ο κόσμος εκεί θα συνεργαζόταν. Έτσι ξεκινήσαμε να πάμε στη Ρουμανία και πρέπει να πω ότι αυτό δεν επαληθεύτηκε καθόλου. Συναντήσαμε ανθρώπους οι οποίοι αρνούν το, αρνούν κατηγορηματικά ότι συνέβη οτιδήποτε στη Ρουμανία. Να σας πω τι κάναμε και στην αποστολή. Πρώτα συναντηθήκαμε με εκπροσώπους Κοινωνία των πολιτών, την Ένωση ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Ρουμανία και με δύο άλλους οργανισμούς και δημοσιογράφους της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Τίποτα δεν είχε προχωρήσει, μας είπαν όλοι αυτοί, ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να φτάσουν σε κάποια πληροφόρηση και αυτό που μας ανησύχησε ήταν ότι αυτή η έρευνα δεν είχε καθόλου τη λαϊκή στήριξη, την υποστήριξη της κοινή γνώμης. Ε, Μετά τις συναντήσεις αυτές ε, είδαμε τον πρώην επικεφαλής των Ρουμανικών Μυστικών Υπηρεσιών και πληροφοριών που ήδη είχε δώσει συνεντεύξεις στο γερμανικό τύπο και είχε παραδεχτεί ότι υπήρχαν κέντρα τέτοια παράνομα στη Ρουμανία κράτησης. Για μας, σε μας δεν ήταν τόσο εύγλωτος ούτε τόσο ξεκάθαρος. Μας είπε ότι βοήθησε ε, τους Αμερικανούς όταν τους ζήτησαν κάποιες εγκαταστάσεις και τους έδωσε τη δυνατότητα πρόσβασης σε κάποιες εγκαταστάσεις αλλά δεν είχε ιδέα τι τις έκαναν τις εγκαταστάσεις αυτές. Και επίση μας είπε ότι δεν είχε ιδέα καν για το πού βρίσκονται αυτές οι εγκαταστάσεις. Μετά τη συνάντηση αυτή, είδαμε ένα εκπρόσωπο του, ε, του Υπουργού Εξωτερικών. Ο πρόεδρος μας, ο κ. Μωράες, είχε στείλει επανειλημμένα επιστολές για να μπορέσουμε να επισκεφθούμε αυτές τις εγκαταστάσεις, ε, τις παράνομες φυλακές που είχαν ε, βρει οι δημοσιογράφοι και οι άλλοι που τις είχαν ανακαλύψει και εντοπίσει. Όνες λέγεται αυτό το μέρος. Αλλά ε, ήταν εδώ ο υπουργό Εξωτερικών και μας δέχτηκε ο, ο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ο οποίος ήταν τελείως αρνητικός και κατηγορηματικός. Αποκλείεται, δεν έχει γίνει τίποτα στη Ρουμανία μας, είπε, παρά τα στοιχεία που είχαμε εμείς στα χέρια μας. Και τα σχόλια του ήταν ότι καλά ακούτε τους δημοσιογράφους τώρα, αυτά είναι αποδείξεις. Με περιφρόνηση για τη δουλειά όλη αυτή των δημοσιογράφων. Μα είπε ότι διεξάγεται έρευνα και εγώ δεν μπορώ να επέμβω στη δικαιοσύνη. Γεγονό είναι αυτό βέβαια, αλλά εμεί το απαντήσαμε ότι εκπροσωπούσε τη χώρα, το κράτο. Και δεν χρειαζόταν ε, την έρευνα αυτή για να γνωρίζει τι γίνεται. Η πολιτική τους είναι να τελείως αρνητικά κλειστή. Ε, ε, όσο δεν μπορεί από την έκθεση να διαβάσει κανείς ότι πρόκειται για τη Ρουμανία, ε, δεν ε, θα ανοίξουν τα χαρτιά τους. Ε, την επόμενη μέρα συναντηθήκαμε με το Γενικό Εισαγγελέα της Ρουμανίας, είναι ο κύριος Τιμπέριου Μιχάη Νίτου, ο οποίος και αυτός κρύφτηκε πίσω από το μυστικό και το απόρριτο της έρευνας, αλλά μας είπε ότι Αποδείξεις δεν είχε καθόλου. Ότι ο κύριος Αλνασίρη, που ξέρετε την υπόθεση αυτή, είναι στο ΕΔΑΔ, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δεν υπήρχε λοιπόν, λέει, καμία απόδειξη ότι είχε κρατηθεί ο κύριος Αλνασίρη στο έδαφος της Ρουμανίας. Καμία. Εγώ αισιόδοξη δεν είμαι πάρα πολύ, προς την έκβαση αυτής της δικαστικής έρευνας. Ε, το ρώτησα πόσους μάρτυρες ε, εξέτασε, σε ποια ακτίνα δηλαδή, πόσο χιλιόμετρων γύρω από την υποτιθέμενη μυστική φυλακή. Από αυτό που μου απάντησε, αποκόμισα την εντύπωση ότι δεν γινόταν πραγματική δικαστική έρευνα. Ε, Και κανένας δεν μπόρεσε να μεταβεί σε αυτό το κέντρο εκεί, το Όνες. Εμείς επιμείναμε πάρα πολύ στη συνεδρίαση με τον Υφυπουργό, αλλά είχε σαφείς υποδείξεις να αρνηθεί. Βεβαίως δεν μας έδωσαν και καμία δικαιολογία για όλα αυτά. Στο τέλος της αποστολής μας είχαμε και μια συνάντηση στο Κοινοβούλιο. Συναντήσαμε τον επικεφαλής της Επιτροπής Αμήνης της Γερουσίας που είναι αρμόδιοι και έκαναν την προηγούμενη έρευνα που είχε αρνητικό αποτέλεσμα και τους ρωτήσαμε εκεί μήπως ξανανοίξει η έρευνα γιατί έχουμε νέα στοιχεία από την έκθεση Feinstein του Δεκεμβρίου 2014. Εκεί στη Γερουσία δεν ήταν τελείως αρνητικοί, έδειξαν κάποια προθυμία να μας ακούσουν, αλλά μας πρότειναν να αποτανθούμε στη γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών για την έκθεση Φάινσταϊν και να μας δώσουν ε, μία ε, μη λογοκριμένη έκδοση της Έκθεση Φάινστάιν. Μα είπαν θα το κάνουν και εκείνοι και έχουμε μάθει στο μεταξύ ότι το ζήτησε. Η γερουσία της Ρουμανίας απετάνθη στην Αμερικανική γερουσία και ζητάει την έκθεση Φάινστάιν χωρίς το λογοκριμένο τμήμα, τη διαγραφή των ονομάτων των κρατών δηλαδή. Αυτά. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε ε, να ερευνούμε το θέμα αυτό και να περιμένουμε και την έκθεση τη μη λογοκριμένη, επαναλαμβάνω, έκδοση της έκθεσης Φάινσταϊν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ζολή, πρόεδρος. προχωρήσουμε τώρα. Ε, στον τελικό μιλητή πρώτα να δώσουμε ε, το λόγο στους ε, ευρωβουλευτές για ερωτήσεις. στην αρχική έρευνα βασιστήκαμε σε μεγάλο βαθμό στον ρόλο ε, ε, δημοσιογράφων ερευνητών. Και τώρα μετά την έκθεση Φάινστάιν θα θέλαμε να ακούσουμε τι έχει να πει ένας από τους δημοσιογράφους αυτούς. Θα δώσω λοιπόν το λόγο ε, στον Κρόφτον Μπλακ. Παρακαλώ. Ναι. Σας ευχαριστώ. Πριν δέκα χρόνια Ακούσαμε την είδηση ότι η CIA είχε μυστικές φυλακές ε, στην Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας ε, είδαμε σιγά σιγά τη σύνθεση ενός παζλ. Ε, εντοπίστηκαν τα κομμάτια, γενικά έχουν τοποθετηθεί στο σωστό μέρος και μεγάλο μέρος της δουλειάς αυτής έχει γίνει από δημοσιογράφους σε διάφορες χώρες, τις Ηνωμένε Πολιτείε, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, τη Γερμανία, το Πακιστάν, την Πολωνία, τη Ρουμανία Πολλή δουλειά έχει γίνει από διεθνείς φορείς, ε, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ε, από την Επιτροπή σας, από μη κυβερνητικές οργανώσεις, από νομικές ομάδες σε όλο τον κόσμο ε, και από αστυνομικές δυνάμεις και εισαγγελίες στην Ισπανία, Πορτογαλία και αλλού. Και πρόσφατα είδαμε την πολλή δουλειά που έχει πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Πληροφοριών της ε, Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, 500 σελίδες ε, με στοιχεία ε, κυρίως από τα αρχεία της CIA. Πολλά είδη δεδομένων έχουν προκύψει από όλη αυτή τη δουλειά. Έχουμε τα ονόματα των ανθρώπων που εξαφανίστηκαν ε, κατά το διάστημα αυτό. Έχουμε ε, καταθέσεις ε, διαφόρων από αυτούς που περιγράφουν πού κρατήθηκαν, πώς τους μεταχειρίστηκαν και ποιοι ήταν οι συγκρατούμενοι τους. Έτσι, έχουμε τις πορείες των πτήσεων, ξέρουμε πού τους πήγανε, ποιες ε, ημερομηνίες, είδαμε πώς έχουν οργανωθεί οι πτήσεις αυτές, ε, ποιος ε, πλήρωσε για αυτές, πόσα χρήματα πληρώθηκαν, έχουμε ένορκες καταθέσεις που δείχνουν ότι οι πτήσεις αυτές είχαν συγκεκριμένο στόχο την μεταγωγή κρατούμενων είδαμε μηχανισμούς ε, κάλυψης ώστε να ε, κρύβουν οι πτήσεις αυτές τον προορισμό τους. Έχουμε επίσης στοιχεία για τον πραγματικό τους προορισμό. Έχουμε ε, μαρτυρίες εργαζομένων στα αεροδρόμια. Έχουμε με λίγα λόγια σχεδόν έναν πλήρη χάρτη του ε, οργανωτικού δικτύου που διευκόλυνε την ε, λειτουργία του προγράμματος αυτού. Και επίσης έχουμε στοιχεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες που επιβεβαιώνουν όλα τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει από άλλες πηγέ. Και θα ήθελα να ε, επιβεβαιώσω αυτήν την, αυτόν τον ρόλο που παίζει αυτή η έκθεση της Γερουσίας, ότι επιβεβαιώνουν δηλαδή τα άλλα στοιχεία. Ε, υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι που έχουν επικεντρωθεί σε ε, κάποια τμήματα της όλης εικόνας. Ε, πολλοί εργάζονταν ανεξάρτητα από τους άλλους, αλλά η έκθεση αυτή επιβεβαιώνει τα προηγούμενα στοιχεία. Ε, η Επιτροπή σας ε, υιοθέτησε ένα ψήφισμα το 2012, έκτοτε έχουν επιβεβαιωθεί τα στοιχεία αυτά και η έκθεση της Γερουσίας επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά τα στοιχεία αυτά. Ε, έχουμε στοιχεία από την Πολωνία από το, το φθινόπωρο του 2012 μέχρι το 2013, στη Ρουμανία από το 2013 ε, 2002-2003 και στην Λιθουανία, στις φυλακές που λειτουργούσαν ε, έχουμε αναλυτικές περιγραφές ε, κάποιων από τα πράγματα που ε, πραγματοποιούνταν εκεί πέρα. Στέρηση ύπνου στο βαθμό να βλέπει κανείς που να έχει κανείς επαρεστήσεις και είναι και άλλα βασανιστήρια και είναι γεγονός ότι κατά διάρκεια αυτή η CIA είχε μια εγκληματική νομοσία στην Ευρώπη και μάλιστα ε, πλήρωνε εκατομμύρια δολάρια στις ε, χώρες ε, που την βοηθούσαν. Αυτό στηρίζεται από πάρα πολλά στοιχεία τα οποία αν τα συνδυάσουμε έχουμε πλήρη ιστορία. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω το ρόλο των δημοσιογράφων ε, στη συλλογή και επιβεβαίωση των στοιχείων αυτών. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ και στην ε, φύση των στοιχείων αυτών ε, και το θέμα της αμφισβήτησης των στοιχείων αυτών, διότι όπως ακούσατε υπάρχουν, υπάρχουν άνθρωποι που τα αμφισβητούν. Οι άνθρωποι που αμφισβητούν τα στοιχεία αυτά αμφισβητούν ε, κυρίως τη διαδικασία με την οποία συλλέχθησαν, την δημοσιογραφία δηλαδή. Ε, υποστηρίζουν ε, ότι δεν μπορούμε να πάρουν στα σοβαρά τα στοιχεία αυτά διότι, έχουν, διότι αποτελούν προϊόν δημοσιογράφων αλλά όπως ακούσατε σήμερα το πρωί δεν είναι ε, βάσιμο το επιχείρημα αυτό ε, και δεν το εφηβρεγό το επιχείρημα αυτό. Ε, διάφοροι αξιωματούχοι στο Ηνωμένο Βασίλειο τα λένε αυτό. Πριν κάποιες εβδομάδες αξιωματούχος από τη Ρουμανία είπε ότι δεν υπάρχουν βάσιμα στοιχεία και αμέσω μετά το Υπουργείο του είπε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να σταματήσει η αναπαραγωγή αβάσιμων ισχυρισμών λοιπόν ε, στο κοινό. Η ισχύση των ε, δεδομένων ε, έχει ήδη γίνει αποδεχτή από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις υποθέσεις Απούζα Παϊδά και Αλνασίρη που αφορούν την Πολωνία. Και το δικαστήριο είπε ότι τα στοιχεία αυτά είναι αναλυτικά, συγκεκριμένα και συνεπή. και ότι ε, αποδείξεις ε, μπορούν να ε, εξαχθούν από τα δεδομένα αυτά. Και στην περίπτωση της Πολωνίας το δικαστήριο είπε ότι είναι αρκετά αξιόπιστα τα στοιχεία αυτά για να θεωρηθούν αποδεικτικά στοιχεία. Εάν δεχτούμε την υπόθεση κατά της Πολωνίας μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι αυτό ισχύει και για τη Ρουμανία και τη Λιθουανία, διότι αυτή είναι η φύση του δικτύου και δεν ε, είναι ασυνήθιστο να συναντούμε ανθρώπους που να λένε ότι ε, λείπουν ε, τα αποδεικτικά στοιχεία. Λένε υπάρχει φωτογραφία των κρατούμενων σε πτήση μεταγωγών ή κάτι τέτοιο. 14.000 τέτοιες φωτογραφίες ανακοινώθηκε ότι υπάρχουν, αλλά πέρα από αυτό θα ήθελα να ε, αναφερθώ στο επιχείρημα ότι μια φωτογραφία θα έκανε τη διαφορά. Και από τη Λιθουανία ακούσαμε παρόμοια επιχειρήματα, παρότι ε, στην περίπτωση αυτή ε, ούτε η φωτογραφία θα αρκούσε, θα έπρεπε ε, να είναι ο Λιθουανός ο ίδιος παρόν είπε ότι δεν ε, κράτησα κανέναν από τους τρομοκράτες από το χέρι. Πώς λοιπόν μπορώ να έχω οριστική απάντηση. Υπάρχει μια ε, ε, γνωστή υπόθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο που αναφέρεται στην βαρύτητα των επιχείρηματων. Θα πρέπει Μπορεί να υπάρχει κάποιος ε, συνδυασμός ε, περιστάσεων ε, όπου η κάθε μεμονωμένη να μην αποδεικνύει τίποτα αλλά εάν τις συνδυάσουμε να μπορούμε να έχουμε σχετική βεβαιότητα. Το γεγονός ότι η CIA είχε φύλακες στην Πολωνία, Ρουμανία και Λιθουανία, ότι είχε κρατούμενος στις χώρες αυτές χωρίς εποπτεία χωρίς ε, δικαίωμα προσφυγής. Ε, ε, νομίζω ότι έχει αποδειχθεί επαρκώς. Θα πρέπει όμως να αναρωτηθούμε γιατί και πώς οι θεσμοί της Ευρώπης που θα έπρεπε να ασχοληθούν με το θέμα αυτό δεν το έκαναν αφήνοντας ένα κενό στη λογοδοσία το οποίο συμπλήρωσαν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, η κοινωνία των πολιτών, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κλπ. δεν νομίζω ότι είναι ε, ανίκανες ε, οι οργανώσεις αυτές, ε, διότι πολύ συχνά έχουν δείξει μεγάλη ικανότητα σε πολύ πιο δύσκολα έργα από ότι το να δείξουν ότι η CIA είχε μυστικές φυλακές στην Ευρώπη. Διότι προσπάθησαν να αποδείξουν το αντίθετο, το οποίο είναι πιο δύσκολο. Ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου είναι πολύ λιγότερο πολύπλοκος από ότι οποιαδήποτε εναλλακτική λύση. Είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο, αδύνατο θα έλεγα, να διατηρήσει ε, να δώσει κανείς νέο νόημα σε όλα τα στοιχεία που τώρα πια υπάρχουν ε, Δηλαδή όλα τα στοιχεία περί πτήσεων, φυλακών, ε, τα περί πληρωμών κλπ. Ε, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να διατηρήσουν όλο αυτό το δίκτυο στοιχείων εάν δεν υπήρχαν οι φυλακές. Υποστηρίχθηκε ότι οι πτήσεις ε, της CIA πήγαν στη Λιθουανία για να μην κάνουν τίποτα. Όσον αφορά το κτίριο, Θεωρείτε ότι μπορεί ε, η CIA να έκτισε τεράστια αποθήκη έξω από το Βίλνιους, ε, μάλιστα με κλιματισμό ε, και πλήρωσε, για να αποθηκεύσει πολύτιμα αντικείμενα και μετά πλήρωσε ένα σωρό πτήσεις που τελικά δεν έφεραν τίποτα στις αποθήκες αυτές. Είναι πολύ δύσκολο να το δεχτεί κανείς αυτό και αν κοιτάξουμε και τις λεπτομέρειες. Θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία δεν απαντώνται καθόλου στην περίπτωση αυτή. για παράδειγμα ότι ε, τα, οι συμβάσεις των αεροπλάνων αυτών βασίζονται σε μια ε, σύμβαση για μεταγωγές και όχι για μεταφορά πολύτιμων αντικειμένων. Ας, ε, ας προχωρήσουμε λοιπόν πέρα από το θέμα αυτό και ας αναρωτηθούμε γιατί οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αρνούνται να ε, ομολογήσουν αυτό που είναι προφανές. Άλλωστε οι ΗΠΑ το έχουν ομολογήσει και ε, έχουν δημοσιεύσει εκατοντάδες σελίδων ε, για το θέμα αυτό. Α αναρωτηθούμε λοιπόν γιατί είναι πιο εύκολο στην Ευρώπη να διατηρεί κανείς μύθους και αντί να ομολογήσει αυτό που όλοι γνωρίζουν ότι είναι αλήθεια. Το θέμα λοιπόν δεν είναι το πότε, πού κλπ λοιπά υπήρχαν οι φυλακές. Το, πραγματικό μυστήριο είναι πώς είναι δυνατόν ε, οι κοινοβουλευτικοί και δικαστικοί μας οργανισμοί να μην αντιμετωπίζουν ε, το θέμα αυτό τώρα που ξέρουμε ότι όλα αυτά συνέβησαν. Thank you very much, Mr. Black. Ευχαριστούμε κύριε Μπλακ. Και τώρα ο λόγος του συναδέλφους που θέλουν ε, να παρέμβουν. Απλώ να πω ότι έχουμε προσκαλέσει και μέλη του Εθνικού Κοινοβουλίου από την Πολωνία, τον Ηνωμένο Βασίλειο και τη Λιθουανία, αλλά δυστυχώ είχαν αλλημένε υποχρεώσει. Και ο πρώην πρόεδρο τη Επιτροπή Εθνική Ασφάλεια και των Υπηρεσιών του Κοινοβουλίου τη Λιθουανία προσφέρθηκε να απαντήσει σε γραπτό ερωτήσει. Κυρία Ζολή, αν θέλετε κάτι να διορθώσετε από αυτά που είπατε στην παρουσίασή σα, με συγχωρείτε, έκανα ένα λάθο. Σας είπα ότι η Transparency International είχε κάνει πάρα πολύ δουλειά για την διερεύνηση του ποιο αεροσκάφος και για πού. Έπρεπε να πω Amnesty International. Η διεθνή Αμνηστία ήταν το σωστό. Συνάδελφοι, έχουμε μόνο 30 λεπτά για τις ερωταπαντήσεις. Γι' αυτό έχω παραμείνει πολύ σύντομα στις εισηγήσεις μου. Παρακαλώ τι δεν κάνετε κι εσείς και με τη σειρά που θα κληθείτε ε, οι συνάδελφοι. Ο κύριος... Κύριος Βόιτ πρώτος. Mr. Voigt, please go ahead. Ε, ναι, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Τώρα έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις. Η Εξεταστική Επιτροπή, από ό,τι φαίνεται, έχει κάνει καταπληκτική δουλειά σε κάποιο βαθμό, αλλά θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα σε αυτό που αφορά τις ΗΠΑ και αυτό που αφορά εμά, του Ευρωπαίου Έτσι δεν είναι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος καταδίκασε τις δραστηριότητες αυτέ και τα βασανιστήρια. Αυτά είναι πολύ ωραία, αλλά παράδεκτο ταυτόχρονα να μην ε, ε, δέχεται να ε, άρει την ασυλία θα πρέπει να το σκεφτούμε εμείς, να δούμε τι θα κάνουμε με τους Αμερικανούς. Όταν λέγουν ότι υπάρχουν εκατοντάδες ε, αποδείξεις, 14.000 φωτογραφίες και λογαριασμοί και τιμολόγια, ε, θα πρέπει ε, ε, να φτάσουμε και σε κάποιους Αμερικανούς, κάποια φυσικά πρόσωπα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να αγγίξουμε αλλά μπορούμε να τους απαγορεύσουμε την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να τους πειράξει κάπως αυτό. Σε ό,τι αφορά τους Ευρωπαίους με την ακύρωση της Συμφωνίας για τον Ασφαλή Λιμένα έχουμε μία νίκη, μία μάχη ε, και δείχνει αυτό ότι δεν κάνουμε εμείς ό,τι θέλουν οι Αμερικανοί αλλά θα πρέπει και οι Αμερικανοί στα πλαίσια διαπραγματεύσεων για συμφωνίες, είτε είναι αυτό το TTIP είτε άλλες συμφωνίες, να κοιτάξουν ε, και να κοιτάξουμε και εμείς κατά πόσο είναι σοβαροί και αξιόπιστη εταίροι για διαπραγματεύσεις και εμπορικοί εταίροι. Αυτό που εμένα με απασχολεί και με ανισχύει είναι τα πέντε κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ε, μπλοκάρουν και δεν θέλουν να συνεργαστούν. Υπάρχει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, δηλαδή μπορεί κάθε Ευρωπαίος να ε, μεταχθεί σε μία από τις πέντε αυτές χώρες όπου ε, μπορεί να συγκαλυφθεί η κράτησή του, ε, να γίνουν βασανιστήρια και με όλες αυτές τις εκατοντάδες αποδείξεις, 14.000 φωτογραφίες, τιμολόγια και αποδείξεις και ονόματα, να μην μπορούμε με το όνομά τους να διώκουμε συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα και να έχουμε και καταδίκες ενδεχομένως. Έχει γίνει τίποτα από αυτές τις πέντε χώρες. Έχουμε ονόματα ανθρώπων που διώκονται. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ. Όχι μόνο έχουμε κάνουμε την έλλειψη λογοδοσία στην Ευρώπη, αλλά και με θύματα βασανιστήριων. Πολλές φορές στην Ευρώπη κιόλας άνθρωποι που πήγαν στο Γκουαντάναμο και ευρωπαϊκές χώρες δέχτηκαν να τους παραλάβουν κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ. Κάποιος που έμεινε 8 χρόνια στο Γκουαντάναμο μετά απελευθερώθηκε και τώρα είναι στην Ουγγαρία λόγω περίεργων ε, συνθήκων και η Ουγγαρία τους δέχτηκε δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν μπορεί να βρει δουλειά, δεν έχει χαρτιά, δεν έχουν χαρτιά ούτε τα παιδιά του και δεν του έχει παρασκευθεί ούτε καν στέγη. Για να μην αναφέρω τις τραυματικές εμπειρίες που έζησε τα 8 χρόνια της κράτησή του και των βασανιστήριων. Έχουμε όμως και πρώην πράκτορες της CIA που επίσης παραπονούνται ότι ήταν θύματα κακής εκδίκασης και δικαστικής πλάνης στην Ευρώπη, συγκεκριμένα στην Ιταλία. Και αυτό βεβαίως έχει χρησιμοποιηθεί ως προκάλημα για να αποκρύψουν του πραγματικού ενόχου στι ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Τι μυστικέ υπηρεσίε που έπαιρναν μέρο σε αυτά τα προγράμματα. όπως η Σαμπίνε Ρεσόζο που ήταν ε, μέλος της CIA, Αμερικανίδα από την Πορτογαλία όμως, η οποία εντοπίστηκε στην Ιταλία και είναι φυσικά εύκολο οι μικροί, οι να την πληρώσουν και να αφαιθούν ελεύθερα, τελεύθερα, ψηλά στελέχη για να συνεχίσουν το έργο τους. Αυτά ως προς τη λογοδοσία. Ήθελα να ρωτήσω και ως απάντηση σε όσα είπε ο κύριος Κρόστον Για όσα είπα για τα αποδεκτικά, με τα αποδεκτικά στοιχεία που έχουμε, με τόσες καταδίκες και με την αντίσταση τόσων ευρωπαϊκών χωρών να απαντήσουν. Λυπούμε που θα το πω. Αλλά είναι τεράστιο θέμα. Και έχει πολύ να κάνει με το πώς οι διαφορετικές κυβερνήσεις ε, αντιλαμβάνονται τις ευθύνες τους και καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους τι βασικέ του υποχρεώσει του, όπω προκύπτουν από το κράτο δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά. Εδώ όμω υπάρχει και μια ευρωπαϊκή προοπτική. Και πρέπει να πω ότι εδώ και μια δεκαετία, διότι αυτό κατάει μια δεκαετία τώρα, ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κ. Ντουράου Μπαρόζο, τη δική μου τη χώρα τη Πορτογαλία, ήταν πρωθυπουργό όταν οι πτήσει και τα βασανιστήρια άρχισαν γίνονται το 2002 και τον οποίο έχω καταγγείλει και έχω ε, υποβάλει αγωγή με συγκεκριμένες κατηγορίες εναντίον του για συνενοχή δεν έχει απαντήσει. Υπάρχουν όλα τα στοιχεία, τα ονόματα, τον, ε, τα στοιχεία που ζήτησα από τον καθηγητή Ντε ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι σύμβουλος παρά το σημερινό πρόεδρο της Πορτογαλίας, για στοιχεία του ευρωπαϊκού δικαίου και για να επιτρέψει ανακρίσεις όχι μόνο σε αεροσκάφη αλλά και σε σκάφη στη θάλασσα. Και βεβαίω υπήρξε τεράστια προσπάθεια συγκάλυψης και από το δικαστικό σύστημα και από την ε, πολιτική έρευνα που θα πρέπει να γίνει στην Πορτογαλία. Τα λέω αυτά, αλλά ήταν και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο κύριος Δουραμπαρόζο. Ε, Ντουραμπαρόζο. Ε, αυτό εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την απροθυμία του να πιέσει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για λογοδοσία και φυσικά ήταν ενεργός, είχε δραστήρια συνενοχή, ενεργό συνενοχή και εκείνος και άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και όλοι προσπαθούν να συγκαλύψουν τις δικές τους ευθύνες. Το ίδιο έκανε και εκείνο από τότε που ανέλαβε πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Η κυρία Κατρίκα. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Η κυρία Κουντρίτσκα. Έχω την εντύπωση ότι στις παρεμβάσεις αυτές που ακούμε κυρίως τις δύο κυρίες που ακούσαμε από το πάνελ. Ε, είναι πολύ μεροληπτικά αυτά που ακούμε και μονομερή. Για ποιο λόγο. Εγώ βλέπω πώς εξελίσσεται η κατάσταση στην Ευρώπη και στα πέντε κράτη-μέλη που εσείς ε, κυρίες μου επικρίνετε. Το 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μάλλον υπήρχε εδώ μια εξεταστική επιτροπή με πρόεδρο τον κύριο Κάρλος Κοέιο που είναι μέλος της επιτροπής μας και έκανε πάρα πολλά για να ευιστοποιήσει την κοινή γνώμη στα λόγω κράτη-μέλη και να ε, ληφθούν ε, τα απαραίτητα μέτρα. Πράγμα που έγινε. Εσείς τι έρχεστε να κάνετε εδώ. Έρχεστε να επικαλεστείτε την απόφαση του δικαστηρίου ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή την έκθεση για τη CIA. Αλλά ε, κάπως ε, παρακάμπτεται τις εξελίξεις στα διάφορα κράτη-μέλη. Δεν τις αναφέρεται. Έρχομαι στην Πολωνία. Λέτε ότι δεν εκτελεί τη δικαστική απόφαση. Μα έχει κάνει έφεση έχει προσβάλει την απόφαση αυτή η Πολωνία, τον Οκτώβριο μάλιστα, πέρσι, για διάφορους λόγους που θα σας αναφέρω. Πρώτον, η πολωνική κυβέρνηση έχει διατάξει κανονική έρευνα ε, μετά τα πορίσματα του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου και τα αιτήματα της πολωνικής κοινή γνώμης. Η έρευνα αυτή κατέληξε με συγκεκριμένα αποτελέσματα κανονικότατα. Ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του 2002, κ. Σινατκόφσκι, ε, διώκεται μετά από την έρευνα αυτή. Το πρόβλημα ποιο είναι. Η πολωνική κυβέρνηση ε, απευθύνθηκε στις Αμερικανικές αρχές για να έχει περισσότερες αποδείξεις. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε να δώσουν στοιχεία εις βάρος τους αυτοί που τότε κυβερνούσαν. Θα πρέπει να απευθυνθούμε σε κάποιον άλλο. Οι Αμερικανοί αρνήθηκαν να μας δώσουν στοιχεία στα πλαίσια της αίτηση δικαστικής συνδρομής μας είπαν ότι δεν θέλουμε να συνεργαστούμε σε αυτό το θέμα με την πολωνική κυβέρνηση ε, για να αποκατασταθούν τα αντικειμενικά γεγονότα ποιος ευθύνεται, γιατί και πότε. Γνωρίζουμε ότι τότε η πολωνική κυβέρνηση ήταν υπεύθυνη για την ύπαρξη χώρων όπου ήταν αυτές οι παράνομες δραστηριότητες και τα βασανιστήρια. Αλλά το θέμα είναι ποιο πήρε την απόφαση. Αυτό είναι, αυτό πρέπει να διερευνηθεί. Και είναι άλλη ιστορία. Επίσης, αποσιωπάται το γεγονό ότι εκτός από την ε, ποινική ευθύνη υπάρχει και η πολιτική ευθύνη. Την πολιτική ευθύνη αναζήτησαν στους επικεφαλείς ε, τότε ε, τους πολιτιακούς ανώτατους παράγοντες, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό. Ε, ήταν σοσιαλιστική, θυμίζω τότε, η κυβέρνηση. Και μετά τα γεγονότα αυτά έχασαν την εξουσία οι σοσιαλιστές και δεν επανήλθαν ποτέ. Το σοσιαλιστικό κόμμα στην Πολωνία είναι πάρα πολύ αδύναμο. Μιλώ λοιπόν για την πολιτική ευθύνη για όλα αυτά τα γεγονότα της εποχής εκείνης. Πιέζουμε λοιπόν από τη μια ε, για να ε, εφαρμόζονται σωστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και από την άλλη να ζητούμε τις πολιτικές ευθύνες των ε, τότε ηθινόντων. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να είστε λίγο πιο ακριβείς στα όσα παρουσιάζετε και λίγο πιο ειλικρινείς δίνοντας αυτές τις πληροφορίες σε ό,τι αφορά την υπόθεση αυτή και πώς τα κράτη-μέλη ανταποκρίνονται και σέβονται τις υποχρεώσεις τους. Αναφέρεται και το άρθρο 38 της Σύμβασης για την ε, διαβίβαση προφοριών και ανταλλαγή. Βεβαίως, υπάρχει αυτό το άρθρο, αλλά δεν υπήρχαν οι πληροφορίε τότε γιατί δεν τις είχαν αποκαλύψει οι Αμερικανοί. Τι θέλετε να διαβιβαστεί, συγγνώμη που σας διακόπτω λέει ο Πρόεδρος, αλλά έχουμε χρονικό πρόβλημα. Για να μιλήσουν όλοι. Η κυρία Νιτφέλτ. Yes, thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μέσα σε λίγες εβδομάδες θα κλείσουμε δεκαετία από τότε που τα πρώτα στοιχεία για τις παράνομες φυλακές και τις παράνομες παραδόσεις και τα βασανιστήρια αποκαλύφθηκαν από τη Washington Post και την Human, Rights Watch. Πριν από 10 χρόνια και πρέπει να πω ότι είμαι περήφανη και ιδιαίτερα ικανοποιημένη που το Κοινοβούλιο διατηρεί το θέμα αυτό προτεραιότητα εδώ και μια δεκαετία. Αλλά πραγματικά είναι ε, απόλυτα θλιβερό που εδώ και δέκα χρόνια δεν υπάρχει παραμικρή λογοδοσία. Καμία λογοδοσία. Σήμερα δημοσιεύεται μια έκθεση στη δική μου τη χώρα, τις κάτω χώρες, για την, ε, για την κατάρριψη του για την, κατάρρυψη για την του MH17 με τρεις θανάτους και καλό θα ήταν με 300 νεκρούς και σημαντικό είναι τουλάχιστον να προσαχθούν οι υπεύθυνοι. Γιατί δεν προχωράει αυτή η υπόθεση. Γιατί. Γιατί μήπως συνεργαστήκαμε με τους ε, δράστες, με τους υπεύθυνους Μήπως είμαστε οι μεσηδράστες, δεν είναι η πραγματικότητα τουλάχιστον ένας από τους πυλώνες του κράτους δικαίου και της δικαιοσύνης. Γιατί δεν ε, υπάρχει λοιπόν λογοδοσία, γιατί δεν επικρατεί το, δεν επιβάλλεται το κράτος δικαίου, γιατί δεν θέτουμε στους εαυτούς μας δυσάρεστες ερωτήσεις. Ένας από τους βασικούς συνεργάτες αυτό το πρόγραμμα ήταν ένας κύριος Ασάντ και η Συρία ήταν ένας από τους βασικούς προορισμούς διότι προφανώς είχαν πολύ καλή μεθόδους ανάκρισης εκεί. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Ασάντ είναι εχθρός μας. Γιατί τις ερωτήσεις αυτές δεν τις θέτουμε, γιατί διαρκώς έχουμε μια αναλυτική αναφορά για το πως ένα μικροσκοπικό κομμάτι του παζλ μπορεί να αποδειχθεί και να ευσταθεί στο δικαστήριο ή όχι. Έχει αποδειχθεί Έχουμε κάνει επανειλημμένους συζητήσει για τις λεπτομέρειες όλων αυτών των θεμάτων. Είναι επιτέλους ε, στιγμή η Ευρώπη να αναλάβει τις ευθύνε της. Και όσοι τα έκαναν αυτά να ε, προσαχθούν σε κάποιο δικαστήριο. Εάν δεν γίνει αυτό, χάνουμε το κύρος μας, το ηθικό μας κύρος, εάν μας έχει μείνει καθόλου. Και χάνουμε και την αξιοπιστία μας. Ελπίζω ότι παρά το γεγονός ότι βλέπω κάποιους εδώ να ε, κάνουν ε, κινήσεις ότι αισθάνονται άβολα σε μια αίθουσα και να κάνουν γκριμάτσες. Εδώ αυτό που θέλουμε είναι η Ευρώπη να αναλάβει ευθύνες και να παραμείνει προτεραιότητα το θέμα αυτό και κάποια στιγμή οι ένοχοι να καταδικαστούν. Ευχαριστούμε κύριε Λόπες Αγγιλάρ. Ευχαριστώ. Να θέσω κάποιες ερωτήσεις στον κύριο Μπλάκ. που εκπροσωπεί τους ερευνητές δημοσιογράφους εδώ και ο καθένας νομίζω μετά από τόσα χρόνια έχει διαμορφώσει τη δική του άποψη μετά τα διαδοχικά βήματα που έγιναν στην Επιτροπή Λίμπερ για τη διαλεύκανση των διαφορών υποθέσεων, για την ε, ανακάλυψη της αλήθειας πίσω από τα διάφορα στοιχεία. Έχει καταλάβει πώς έχουν παραβιαστεί τα θεμελιώδη δικαιώματα και σίγουρα θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί. Υπάρχουν όμως κάποια συγκεκριμένα σημεία όπου νομίζω ότι η δική σας μαρτυρία μπορούσε πραγματικά να μας διαφωτίσει. Πρώτα-πρώτα, μετά από όλες τις έρευνες που έχουν γίνει, ήθελα να μου πείτε τι γνωρίζετε για τους κρατουμένους, αυτούς που έχουν υποφέρει από τις ε, κακές μεθόδους και τα βασανιστήρια και που μπορεί να μην είχαν καμία σχέση με την τρομοκρατία, καμία σχέση με τρομοκρατικές ενέργειες ή εγκλήματα. Καμία σχέση λοιπόν με τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας που ε, υποθετικά ήταν ε, το αίτιο όλων αυτών. Έπειτα, το άλλο που θέλω να μου πείτε αν γνωρίζετε είναι κατά πόσον υπήρχε κάποια συμφωνία που συμπεριελάμβανε ή υπονοούσε ότι θα υπάρχει κάποιο είδους αμοιβή για όσους εμπλέκονταν στην όλη υπόθεση. για τους ε, συνεργούς όλων αυτών των περιπτώσεων. Κάποιο είδους δωροδικία, κάποιο είδους οικονομική αμοιβή ή κάτι τέτοιου είδους. Και η τρίτη ερώτηση είναι τι γνωρίζετε για το επίπεδο λογοδοσίας που έχει καταρτιστεί, διότι όλοι μπορούμε να υποθέσουμε ότι ακόμα και σε χώρες που έχουν εμπλακεί σε τέτοιου είδου ε, πρακτικές και μάλιστα στα υψηλότατα ε, επίπεδα κλιμάκια. Κανείς λέει δεν το γνώριζε. Πώς γίνεται. Ε, πόσο γνωστό ήταν. Μόνο οι μυστικές υπηρεσίες γνώριζαν. Οι υπουργοί. Υπουργοί εξωτερικών, υπουργοί Αμυνα, οι συνεργάτες των πρωθυπουργών. Το επίπεδο λοιπόν αυτό γνώσης, πού φτάνει και ποια είναι η δική σας αξιολόγηση της κατάστασης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κοέλιου. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ τους ομιλητές μας. Έχω κάποιες ερωτήσεις και εγώ. Μάλλον δεν έχω ερωτήσεις να θέσω, αλλά έχω να πω ένα-δύο πράγματα. Πρώτον, να θυμίσω πως όλα ξεκίνησαν στο κοινοβούλιο εδώ. Αρχικώς κάποιοι δεν πίστευαν απλώς ο, τις διάφορες κατηγορίες. Όλοι έλεγαν ότι σε δημοκρατικά κράτη επικρατεί το κράτος δικαίου, το ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν γίνει τέτοια πράγματα. Κατά τη διάρκεια της έκτακτης επιτροπής μας, είδαμε ο ίδιος ο Τζορτ Μπούς σε μία δήλωσή του να αναγνωρίζει τα πάντα εκτός από τα βασανιστήρια. Αναγνώρισε τις παραδόσεις, τις μυστικές φυλακές και ούτω καθεξής. Τώρα έχουμε μία έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ όπου αναγνωρίζει η έκθεση ότι πραγματοποιήθηκαν βασανιστήρια. Δεν μιλούμε πλέον για εικασίες, μιλούμε για γεγονότα και επ' αυτών πρέπει να εργαστούμε. Στην Πορτογαλία λέμε ότι το λάδι ανεβαίνει πάντοτε πάνω σε ένα ποτήρι που έχει και νερό. Και έτσι πιστεύουμε και για αυτή την περίπτωση ότι κάποια στιγμή ο καρπός θα οριμάσει και θα πέσει. Αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε απαθιστό χρόνο. Πρέπει να δουλέψουμε κι εμείς. Γι' αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς Πρόεδρε και την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και όλους όσοι συνεργάζονται μαζί μας που κάνετε σωστά τη δουλειά σας. Διότι δεν μπορούμε να περιμένουμε την ιστορία. Όχι μόνο γιατί πρέπει να υπάρξει ένα αποτέλεσμα, αλλά γιατί προτού υπάρξει το αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τα ίδια πράγματα να ξανασυμβαίνουν. Και πολλοί το επιθυμούν αυτό. Είμαι κυβερνητικέ οργανώσει, να θυμίσω την Διεθνή Αμνηστία και την ε, Human Rights Watch, ο τύπο, οι εθνικέ αρχέ, μεταξύ των οποίων οι δικαστικέ αρχέ, και εδώ να τονίσω την εξαιρετική δουλειά του δικαστού Σπατάρο στην Ιταλία, και βεβαίως το Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι στις μέρες μας κανείς στην Επιτροπή μας δεν μπορεί να αρνηθεί ότι συνέβησαν όλα αυτά και θα πρέπει βάσει αυτής της ε, παραδοχής να εργαστούμε. Θα συμφωνήσω με τη Σοφή που είπε πριν από λίγα λεπτά ότι Θα πρέπει να προτείνουμε λύσεις, θα πρέπει οι ένοχοι να δικαστούν αλλά θα πρέπει και σε πολιτικό επίπεδο να κάνουμε τη δουλειά μας. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε. Νομίζω ότι δύο πρέπει να κάνουμε πρώτα. Δύο τι να. Πρώτα απ' όλα να μην εγκαταλείψουμε την ελεύθερη τη συζήτηση σε επίπεδο Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Θα πρέπει να συνεχίσουμε και να τα φέρουμε και εις πέρας. Αλλά θα πρέπει να παραμείνουμε πιστοί στα γεγονότα. Το κοινοβούλιο αυτό έχει εγκρίνει πολλές χειροπιαστές συγκεκριμένε συστάσεις προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, προς τα κατημέλη, τα διεθνή θεσμικά όργανα. Νομίζω ότι πρέπει επιτέλους να ε, ε, δούμε κατά πόσο οι συστάσεις μας παρακολουθούνται και ακολουθούνται ή όχι. Εάν δεν ακολουθούνται, γιατί συμβαίνει αυτό. Η ερώτηση, η βασική λοιπόν είναι το γιατί. Εάν απαντήσουμε σε αυτό το γιατί, μάλλον θα έχουμε και πολλές σαφείς εξηγήσεις για πολλά θέματα και για πολλούς. Ευχαριστούμε η κυρία Μανέσκου. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω λίγες παρατηρήσεις για την αποστολή της αντιπροσωπείας της ΛΥΠΕ στο Κουρέστι. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι οι αρχές της Ρουμανίας επικρότησαν ε, την επίσκεψή μας, καλωσόρισαν και αυτό φάνηκε από ε, την ε, διοργάνωση των διαφορών συναντήσεων, εκτός από τη συνάντηση με τον Υπουργό, ο οποίος βρίσκονταν στις Βρυξέλλες τότε και με τον κύριο Ηλιέσκου, τον πρώην Πρόεδρο, τον οποίον δεν μπορέσαμε να συναντήσουμε. Όλοι, όλες οι άλλες αρχές συναντήθηκαν με την αντιπροσωπεία μας ε, και αυτό ήταν θετικό δείγμα ότι οι αρχές της Ρουμανίας θέλουν να διατηρήσουν το διάλογο. Ε, η Ρουμανία είναι μέλος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και έχει υπογράψει την σύμβαση κατά των βασανιστήριων ε, και είναι απόλυτα αφοσιωμένη στις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να εργαζόμαστε με την θεωρώντας ότι οι Ρουμανικές αρχές ε, γνώριζαν ε, την ύπαρξη των ε, κέντρων κράτησης και το αποσιωπούσαν. Θα πρέπει να γνωρίζουμε τα, την πραγματικότητα και σε έκθεσή της η γερουσία της ε, Ρουμανίας ε, ε, έλεγε ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη κέντρων κράτησης στη Ρουμανία. Στην έκθεση της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών δεν αναφέρεται η Ρουμανία, συνεχίζει όμως να υπάρχει ο ισχυρισμός και νομίζω ότι είναι προς συμφέρον δικό μας και της Ρουμανίας να ανακαλύψουμε ποια είναι η αλήθεια, διότι το να συνεχίζονται αυτές οι κατηγορίες ε, δεν ωφελεί κανέναν. Πρέπει να γνωρίζουμε την αλήθεια και γι' αυτό στη Ρουμανία αυτή τη στιγμή ε, ε, έχουμε μια ανοιχτή δικαστική διαδικασία για το θέμα αυτό. Συναντηθήκατε με τον Γενικό Εισαγγελέα. Θέλουμε λοιπόν απόλυτη διαφάνεια αλλά βέβαια σεβόμενοι τα όσα μπορούν να επιτρέπεται να υποθούν κατά τη διάρκεια μιας ε, ανοιχτής υπόθεσης. Όσον αφορά λοιπόν ε, την ε, λογοδοσία αλλά και την διάθεση των αρχών να συνομιλήσουν μαζί μας, θα πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη, διότι δεν θέλουμε να κατηγορήσουμε κάποιον άδικα, θέλουμε να ανακαλύψουμε ποια είναι αλήθεια. Χρειάζεται λοιπόν ισορροπία σε όλα όσα κάνουμε. Όσον αφορά τις έρευνες που μας παρουσιάσατε, είναι πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία αυτά. Θεωρείτε εξ αρχής ότι έχετε αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία όμως δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα. Προτιμάμε λοιπόν να στηρίξουμε τις αρχές της Ρουμανίας στην ε, δικαστική υπόθεση, να τις υποστηρίξουμε και όχι απλά να τις κατηγορούμε και να ανακαλύψουμε εάν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος στη Ρουμανία. Εάν ναι, τότε θα πρέπει να καταδικαστεί. Μέχρι τότε όμως θέλω να είμαστε ειλικρινείς και να βλέπουμε τα γεγονότα ως έχουν διότι θα ήθελα να επαναλάβω ότι στην έκθεση της Αμερικανικής ε, Γερουσίας δεν αναφέρεται πουθενά η Ρουμανία. Θα με ενδιέφερε ε, να δω εγώ ίδια τα αποδεικτικά στοιχεία. Ευχαριστώ. Ναι. Θα δώσω το χρόνο για να απαντήσουν οι ομιλητές μας τελευταία ομιλήτρια, η κυρία Παγάσα Ορτοντούα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ απολύτως και με την κυρία Ενετφέλτ και με τον κύριο Κοέγιο. Η ατιμορρυσία θα ήταν ό,τι χειρότερο. Διότι αυτή θα αποδυνάμωνε την ε, αξιοπιστία των θεσμικών μας οργάνων και τις αξίες. Ε, δεν πρέπει να είμαστε ε, και δειλή. Αφού το φτάσαμε ως εδώ μετά από 10 χρόνια θα πρέπει να συνεχίσουμε. Καλή είναι η πολιτική δουλειά και οι συστάσεις, αλλά χρειάζεται και συνέχεια. Και έχω και μια ερώτηση. Σε αυτό το διάλογο με τους ομολόγους μας, ε, των Ηνωμένων Πολιτειών σκεφτόμαστε να κάνουμε καμία αποστολή εμείς στις Ηνωμένες Πολιτείες ως Επιτροπή για να τα μάθουμε από πρώτο χέρι. Ρωτάω επειδή είμαι καινούρια, μπορεί να το έχετε ήδη κάνει. Εγώ θέλω να εθαρρύνω και να συγχαρώ τους συναδέλφους που έχουν παραμείνει στην αναζήτηση της αλήθειας όλα αυτά τα χρόνια, μια δεκαετία ολόκληρη. Ε, πραγματικά πρέπει να είμαστε γνήσιοι εδώ και όχι δίθεν σε αυτή την προσπάθεια, ούτε να ε, είμαστε ητοπαθείς. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο τώρα για να απαντήσουν οι ομιλητές μας από το πάνελ. Ξέρετε ότι από χρόνο δεν πάμε καθόλου καλά, αλλά είναι πολύ σημαντικό οι συνάδελφοι να έχουν την ευκαιρία να... και την ελευθερία να πούν αυτό που θέλουν να πούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να ενημερωθούμε ε, και να επαναλάβουμε τα όσα είχαμε πει το τελευταίο διάστημα, γιατί έχουμε και νέους βουλευτές. Λοιπόν, Πέντε λεπτά, το ξέρω ότι δεν είναι αρκετά για να απαντήσετε. Θα μιλήσει μία από τις δυο σας από το κέντρο το δικό σας, κύριε Αγγελ, κύριε Δαντέσκου και κύριος Πλακ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, και ευχαριστώ όλους τους ομιλητές για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις σας. Δύο συγκεκριμένες παρατηρήσεις θα ήθελα να αντιτάξω σε κάποιες από τις επικρίσεις της έκθεσης. Η πρώτη είναι, είμαστε δίκαιοι απέναντι στα κράτη-μέλη που ε, κατηγορήθηκαν. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα από τα αποδεκτικά στοιχεία που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θεώρησε χρήσιμο να συμπεριλάβει στην ε, απόφασή του για τον Αλ Και αυτό είναι πώς η CIA βρήκε την υπηρεσία πληροφοριών στην Πολωνία με την οποία συνομίλησε και συμφώνησε ε, τη δημιουργία των ε, φυλακών, την διακπαιδεύση των πτήσεων κλπ το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θεώρησε ενδιαφέρον να συμπεριλάβει στην απόφαση ότι το CIA επέλεξε ε, την στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών ε, της Πολωνίας, διότι ήταν η μόνη υπηρεσία της Πολωνίας ε, χωρίς δημοκρατική λογοδοσία. Νομίζω ότι αυτό είναι ενδεικτικό των προβλημάτων που έχουμε με τη δημοκρατία. Αυτό συνδέεται με μια άλλη έκθεση που είχαμε ε, εκπονήσει για σας που έχει να κάνει με την εποπτεία των ε, υπηρεσιών πληροφοριών. Όταν ε, ένας σημαντικός και ισχυρός σύμμαχος θέλει να υπονομεύσει την δημοκρατική λογοδοσία θα πρέπει να αντιστεκόμαστε. Η δεύτερη παρατήρησή μου ε, αναφέρεται σε ένα παράδειγμα 20 ετίας. Υπήρχε ένα πρόβλημα με ε, Υπουργείο Εταιρικών ενός ε, κράτους μέλους σε σχέση με μια τρομακρατική απειλή. Μια ομάδα εντός ενός δημοκρατικού κράτους επέτρεψε σε τάγμα θανάτου ε, να κινητοποιηθεί εντός κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ε, έγινε γνωστό δημοσίως, ε, άλλαξε η κυβέρνηση, έχασε την εξουσία η σοσιαλιστική κυβέρνηση και ο εισαγγελέα κατηγόρησε συγκεκριμένα άτομα συμπεριλαμβανομένου του Υπουργού Εσωτερικών που ήταν υπεύθυνο παρότι ισχυριζόταν ότι δεν είχε γνώση του θέματος. Πολλοί πήγανε φυλακή συμπεριλαμβανομένου του Υπουργού Εσωτερικών. Η χώρα αυτή είναι αφοσιωμένη στη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Ελσπετ, θα μπορούσαμε να είχαμε ακούσει πολύ περισσότερα από την Ελσπετ. Θα ήθελα όμως να την ευχαριστήσω πολύ για την ε, έκθεση της και την δουλειά που έχει κάνει, καθώς να την ευχαριστήσω και για την προηγούμενη δουλειά της ε, για την Επιτροπή μας. Να ακούσουμε την Εύα Ζολή. Παρακαλώ. Well. Λοιπόν, πώς να το πω. Εμείς ε, βεβαίως αποτείουμε φόρο τιμής και τιμούμε και Εκτιμούμε το γεγονός ότι μας δέχτηκαν οι Ρουμανικές Αρχές. Ο Υπουργός Εξωτερικών δεν μπόρεσε να μας δεχτεί διότι ήταν στις Βρυξέλλες, το είπα προηγουμένως και αυτό. Αλλά δεν μπορώ να κρύψω ότι με ενόχλησε πάρα πολύ το γεγονός ότι εκείνοι με τους οποίους συνομιλήσαμε δεν εξέτασαν καν τις αποδείξεις που έχουν συλλεγεί εδώ και δέκα χρόνια από τόσους πολλούς. Και αυτά τα στοιχεία ε, ε, εντυπωσιάζουν τον οποιοδήποτε ασχοληθεί μαζί τους και τα κοιτάξει για 10 λεπτά. Το ξέρω ε, ότι η έκθεση Feinstein δεν κατονομάζει κανέναν. Αλλά εκείνοι το αρνούνται. Για λόγους που εσφαλμένα θεωρούν ότι είναι κάποιοι σύμμαχοί τους που έχουν κάνει μυστικές συμφωνίες με τους Αμερικανούς, αλλά δεν έχουν καταλάβει ακόμα ότι η μυστική συμφωνία έχει σπάσει από την πλευρά των Αμερικανών και δεν έχει νόημα να τους καλύπτουν. Τώρα μπορούν να μιλήσουν. Και θα καλούσα όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου που δεν έχουν πιστεί από την ισχύ των αποδείξεων και που νομίζουν ότι μπορούν να τις κάνουν έτσι στην άκρη. Να το διαβάσουν. Καθηγητές θα έχουν φέρει υπόψη μας και δημοσιογράφοι που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους για τη δική μας ασφάλεια και τη δημοκρατία. Αν θέλετε μπορώ να συγκαλέσω μια συνεδρίαση και να σας καλέσω σας κυρία Μανέσκου για να ε, έρθετε με τον κύριο Μπλακ να σας δείξουμε κι εγώ ε, όλους τους ισχυρισμούς και τις εικασίες που σταμάτησαν στο Βουκουρέστι από, ε, ας πούμε, και για όλες τις πτήσεις. Μαρόκο, Καμπούλ, μέσω Βουκουρεστίου. Και σταμάτησαν στο Βουκουρέστι οι πτήσεις αυτές. Για ποιο λόγο. Παρακαλώ να μην παγιδευτείτε σε αυτή την επιχείρηση συγκάλυψης. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν ε, συνοπτικοί και συγκεκριμένοι. Θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι συνοπτικός. Μόνο μερικές παρατηρήσεις. Πρώτον, σε ό,τι αφορά το κατά πόσο στην Πολωνία οι αρχές παραγωνίστηκαν διότι δεν απαντήσαν οι Ηνωμένε Πολιτείε στο αίτημά τους για συνδρομή ναι, υπήρξε έτοιμα για συνδρομή, όμω νομίζω ότι η Πολωνία έχει ήδη στα χέρια τη όλε τι πληροφορίε που χρειάζεται. Νομίζω ότι είναι και λογικό και ορθό καθώς η Πολωνία έχει αποδείξει με τις δράσεις των μυστικών της υπηρεσιών και υπάρχει απόρριτο φάκελο στα χέρια του εισαγγελέα, εφόσον έχουν τέτοια στοιχεία, γιατί πρέπει αυτός ο φάκελος να κλείσει. Νομίζω ότι οι πληροφορίε στην Πολωνία είναι αρκετέ για να διεξαγάγουν τη δική του έρευνα χωρί να υπολογίζουν στη βοήθεια των ΗΠΑ που μπορεί να μην έρθει και ποτέ. Στι ερωτήσει επί των λεπτομεριών, όπω του κυρίου Λόπε Αγγιλάρ, για τον αριθμό των ατόμων που κρατήθηκαν σε παράνομε φυλακέ που δεν είχαν καμία σχέση με τρομοκρατικέ ενέργειε υπό μία έννοια. Είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς ακριβώ αυτή την ερώτηση. Διότι η έκθεση τη Αμερικανική Γερουσία αναφέρει τουλάχιστον 26 τέτοια άτομα βάσει του ορισμού τη ίδια τη. CIA αλλά κατά πρώτον δεν ξέρουμε εάν ο ορισμό τη. CIA ήταν ο ίδιος σε κάθε περίπτωση και έπειτα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι από του 118 άνθρωπους που ονομάζονται στην, κατονομάζονται στην έκθεση αυτή, ένα τρίτο έχουν σβηστεί από τα αρχαία ούτως ή άλλως, οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε καν για αυτούς. Η έκθεση βέβαια είναι απλώς μία περίληψη. Είναι η ψηροπτική εικόνα μιας ε, απόρριτης έκθεσης 6.000 σελίδων. Και νομίζω ότι υπάρχει ένα κεφάλαιο, ένα υποκεφάλαιο ε, ανά άτομο σε κάθε περίπτωση. Αλλά αυτό δεν το έχουμε στην περίληψη, έχουμε απλώς το κατάλογο. Ένας από τους ανθρώπους που κρατήθηκε ξύπνιος επί σειρά ημερών μετά από αυτή, και έφτασε σε κατάσταση παρεστήσεων τρόμου ήταν ένας άνθρωπος που ονομάζεται Τζόναθαν Κου, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση βάσει των υποψιών της CIA με δημοκρατικές ενέργειες και γι' αυτό και τον απελευθέρωσαν. Κάνατε ερωτήσει που είναι δύσκολο να απαντηθούν. Σε κάθε περίπτωση δεν ξέρουμε σε κάθε χώρα το επίπεδο και το βαθμό στον οποίο στελέχη και κλιμάκια ήταν ενημερωμένα, ποιο γνώριζε και ποιο ακριβώς όχι. στην Πολωνία, ο τότε Πρωθυπουργό και Πρόεδρο μάλλον έχουν αναγνωρίσει ότι τα γνώριζαν στη Ρουμανία. Είδαμε ότι υπήρξε εν μέρη παραδοχή, αλλά υπήρξε και προστοδρόμηση. Η παναχώρηση μάλλον ε, στη Λιθουανία. Ο πρόεδρο Αντάμισκου είπε ότι δεν γνώριζε τίποτα αλλά από την έκθεση της Γερουσίας φαίνεται ε, ότι αρκετοί επίσημοι γνώριζαν στις περισσότερες περιπτώσεις. Υπήρχαν συνομιλίες μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ και των ε, ομόλογων Υπουργείων στην Ευρωπαϊκή Κράτη που ε, δείχνουν ότι γίνονταν συνεννοήσεις. Δεν υπάρχει λοιπόν περίπτωση να μην γνώριζε κανείς. Και όσο για τις ερωτήσεις σας για τα χρηματικά ποσά, υπάρχει ένδειξη από την έκθεση ότι η Ρουμανία έλαβε 8 εκατομμύρια δολάρια λόγω χάρη για αυτή την υπόθεση. Δεν ξέρουμε τι ποσά δόθηκαν στις υπόλοιπες χώρες, αλλά φήμες υπήρξαν ότι σε μια περίπτωση υπήρξαν τεράστιο χαρτοκιβώτιο με χαρτονομίσματα. Η CIA το θεώρησε, το ονόμασε αυτό επιδότηση για τη συνεργασία τους, μπορεί να το πει κανείς δωράκι, πείτε το πως θέλετε. Και μια τελική παρατήρηση. Μπορούμε να, να παραξανευόμαστε, να διαρωτόμαστε τι ακριβώς σημαίνει απόδειξη, ο όρος αυτός, αποδεκτικό στοιχείο, όμως εν τέλει δεν υπάρχει καμία ε, ε, κανένα ίχνος απόδειξης ότι η φυλακή που η έκθεση της CIA αναφέρει ως παράνομη δεν βρισκόταν στη Ρουμανία. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να βρισκόταν κάπου αλλού. Εάν δείτε τις συμβάσεις, τις αποδείξεις, τα τιμολόγια, ε, την εκμίσθωση, τα πάντα και προσπάθησα να το καταστήσω σαφές στην παρουσίασή μου σήμερα, εάν τα δείτε όλα αυτά θα πρέπει κανείς να ε, φανταστεί και να χτίσει ένα φανταστικό παράλληλο κόσμο για να πιστέψει ότι όλα αυτά δεν συνέβησαν στις χώρες που ονομάσαμε. Και σίγουρα αυτό που ε, αναφέρθηκε για την παράνομη φυλακή ήταν σίγουρα στη Ρουμανία και αυτό είναι πέραν κάθε λογικής αμφιβολίας ε, αληθινό. Ευχαριστούμε κύριε Μπλακ, ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες στο πάνελ για τις εξαιρετικές τους συνεισφορές. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Να πάμε κατευθείαν στο επόμενο σύνολο εμπειρογνωμονών, το επόμενο πάνελ. Ο κύριος Ντάφη δεν μπορεί να είναι σήμερα μαζί μα δυστυχώ. αλλά θα ζητήσω... η κυρία Ντάφη δεν μπορεί να είναι σήμερα μαζί μα. θα ζητήσω από του υπόλοιπου να έρθουν ε, στο βήμα. Και επειδή είπαμε και για του ενδιαφερομένους, να ευχαριστήσω και τι μη κυβερνητικέ οργανώσει που συμμετείχαν ήδη από την αρχική έρευνα την Διεθνή Αμνηστία, την ε, Open Society και όλους για τις πρωτοβουλίες τους. Um, Συνάδελφοι, θα προχωρήσουμε τώρα στο δεύτερο πάνελ. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον πρώτο μας ε, προσκεκλημένο, τον κύριο Αρμάντο Πατάρο, που αυτή τη στιγμή είναι ε, εισαγγελέα στο Τωρίνο και είναι γνωστός για την καταδίκη 23 Αμερικανών ε, για την απαγωγή του Αμπού Ομάρ. Καλώς ήρθατε, παρακαλώ. Grazie. Ευχαριστώ. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ και χαίρομαι που βρίσκομαι για άλλη μια φορά στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχω στη διάθεσή μου 15 λεπτά. Αυτό μου επιβάλλει να κάνω κάποιες επιλογές για το ποια θέματα ακριβώς θα θίξω τα άλλα, την υπόθεση της απαγωγής ε, του Αμπού Ομάρ την έχω αναπτύξει πολλές φορές στο Κοινοβούλιο, τη γνωρίζετε. Και στην περίπτωση που προέδρευε στην έκτακτη επιτροπή ο κύριος Κοέλιου. Και εφόσον χρειαστεί μπορώ να σας στείλω και γραπτές, ε, γραπτά στοιχεία για τις εξελίξεις που έχουν προκύψει. Συνοπτικά, να πω απλώς πώς ολοκληρώθηκε η υπόθεση αυτή. Υπάρχουν και κάποια μικρά σφάλματα στην εξαιρετική έκθεση που εκπονήθηκε από την Επιτροπή Λιμπέ. Οι Αμερικανοί που τελικώς καταδικάστηκαν δεν ήταν 22 μέλη της CIA και ένας επιπλέον, αλλά 26 υπήρξε μια δεύτερη απόφαση που οδήγησε σε συνολικό αριθμό 26 τους Αμερικανούς που τελικώς καταδικάστηκαν, 5 ήταν διπλωμάτες. Το δικαστήριο βάσει της δικής μας τοποθέτησης απέριψε την ε, άσκηση της διπλωματικής ασυλίας και έτσι καταδικάστηκαν. Καταδικάστηκε και ένας Ιταλός, ένας χωροφύλακας, ο οποίος ε, ομολόγησε ότι συμμετείχε με ενεργά στην απαγωγή. Δύο ε, από τις μυστικές υπηρεσίες και ένας δημοσιογράφος επίσης καταδικάστηκαν καταδικάστηκαν για διευκόλυνση. Και για τους Ιταλούς μέλη των μυστικών υπηρεσιών υπήρξαν πολλές διαφορετικές αποφάσεις ε, που ήταν αντιφατικές μεταξύ τους, αλλά τελικώς το εφετικό δικαστήριο του Μιλάνου τους καταδίκασε. Ο αρχηγός των υπηρεσιών στη σοβαρότερη τιμωρία, πέντε καταδικάστηκαν, αλλά για το κρατικό μυστικό που μια άλλη κυβέρνηση επικαλέστηκε και τα λέω τώρα κάπως συνοπτικά το συνταγματικό δικαστήριο θεώρησε ότι η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ασκηθεί και το ακυρωτικό δικαστήριο τελικώς απέρριψε και την απόφαση του συνταγματικού. Αλλά να τα δούμε με τη σειρά. Υπάρχει εδώ έλλειψη ισορροπία προφανώ μεταξύ των 26 Αμερικανών, των οποίων η καταδίκη είναι οριστική και τελεσίδικη, και των ε, ε, υπαλλήλων του ΣΥΣΜΗ, των μυστικών υπηρεσιών που έχουν κατηγορηθεί για συνενοχή και οι οποίοι δεν ε, θωώθηκαν. Δεν μπόρεσε να θεωρηθεί ότι ισχύει εδώ το κρατικό μυστικό. Θέλησα λοιπόν να μιλήσω για το κρατικό απόρριτο όπως ορίζεται στη δική μας νομοθεσία αλλά νομίζω ότι αυτά ισχύουν για όλους διότι η περίληψη της παρουσίασής μου είναι αυτή, η ουσία της παρουσίασής μου είναι αυτή. Δεν είναι ότι είναι αδικαιολόγητο και αβάσιμο το κρατικό απόρριτο. Ακόμη και σε δημοκρατική καθεστώτα υπάρχει ανάγκη να ε, εξασφαλίζεται απόρριτο για την προστασία των πολιτών. Το πρόβλημα είναι η κατάχρηση αυτού του απορρίτου και η έλλειψη του πολιτικού ελέγχου. Ε, στην περίπτωση της Ιταλίας πολλές φορές και δικαστικού ελέγχου. Έτσι, ο Ευρωπαίος πολίτης, όπως θα και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, περιμένει όλα αυτά να ελεγχθούν. Να θυμίσω ότι ο Αμπού, ο Μαρκέ εκείνος, καταδικάστηκε για τρομοκρατικές ενέργειες σε έξι χρόνια κάθερξη. Εάν δεν είχε απαχθεί, θα βρισκόταν στη φυλακή με τους ενεργούς του. και μάλιστα μάλλον θα έχει εκτίσει και την ποινή του. Ε, συνολικά, όπως είπα, το κρατικό απόρριτο μπορεί λοιπόν να εφταθεί νομικό σε δημοδιωτικά καθεστώτα. Απλώς πρέπει να βρεθεί ένα σωστό σημείο ισορροπίας μεταξύ των απαιτήσεων της δικαιοσύνης, που πρέπει να βεβαιωθεί ότι αναλαμβάνει τι ευθύνε τη και τι ανάγκε ασφάλειας για τι οποίε έχει προβλεφθεί το κρατικό απόρριτο. Όταν λοιπόν σε μια δικαστική έρευνα προκύπτει το κρατικό απόρριτο, είναι, δημιουργείται μια κατάσταση έντασης μεταξύ της εκτελεστικής εξουσίας και της δικαστικής. Στην Ιταλία υπάρχει ένας νόμος ιδιαίτερα ιδιαίτερα ε, συνεκτικός, ο οποίος εγκρίθηκε το 2007 με αφορμή την υπόθεση του Αμπού Ομάρ. Δύο φορές εμπλέκονται εδώ, δύο οργανισμοί που ονομάζονται υπηρεσίες, κατά στην Ιταλία πολλές φορές αλλάζουν τα ονόματα των οργανισμών, των δημόσιων φορέων, κάποιες φορές λοιπόν ονομάζονται υπηρεσίες και υπάρχει εδώ συγκεκριμένη αρμοδιότητα ε, που έχει να κάνει με το κρατικό απόρριτο και την οποία επικαλείται και επιβάλλει ο Υπουργό Εσωτερικών. Μπορεί να αφορά έγγραφα πληροφορίες, δραστηριότητες των οποίων η διάδοση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην ακυρεότητα τη δημοκρατία ω προ τι διεθνεί συμβάσει που έχει συνάψει ή την υπεράσπιση των φορέων που ε, προβλέπονται από το Σύνταγμα, την ανεξαρτησία του κράτου σε σχέση με άλλα κράτη, την ε, άμυνα και την στρατιωτική ασφάλεια του εν λόγω κράτου. Έτσι ασκείται το κρατικό απόρριτο. Εδώ λοιπόν μια δυνατή συμφωνία μπορεί να ε, ανακληθεί ε, και να υπάρξει ανάλογη συνεννόηση με τα κράτη που έχουν συμβληθεί στην ίδια συμφωνία. Η Ιταλία λοιπόν έχει αυτόν τον υπέροχο νόμο για το, για το κρατικό απόρριτο, το οποίο, ε, το οποίο το πεδίο έχει διευρυνθεί με άλλε δευτερογενεί αποφάσει. Σκεφτείτε μετά από το νόμο του 2007 να εγκρίνεται από το Κοινοβούλιο ότι το κρατικό απόρριτο μπορεί να αφορά και οικονομικά συμφέροντα. Όμω, ο, κ. Πρόντι με την πρωθυπουργικό διάταγμα ε, ε, διευρύνει και άλλο το κρατικό απόρριτο με τα οικονομικά συμφέροντα. Ο νόμος λοιπόν, ο κρατικός νόμος που έχει εγκριθεί από το Κοινοβούλιο ε, έχει αποκλείσει τα οικονομικά συμφέροντα από το κρατικό απόρριτο, ενώ ο κ. Πρόντι τελικά το εισάγει. Αυτό που βγήκε από την πόρτα, λοιπόν, μπαίνει από το παράθυρο. Είναι σημαντική στην περίπτωση αυτή προφανώς ο έλεγχος. Έχουμε δύο ειδών ελέγχους στην Ιταλία, τον πολιτικό και τον δικαστικό των ε, πολιτικών τον αναλαμβάνει μια κοινοβουλευτική επιτροπή κατά πλειοψηφία με μέλη της κυβέρνησης του κυβερνώντος σχηματισμού και ε, με συμμετοχή μελών της αντιπολίτευσης του οποίου το ακρόνιμο είναι κόπεσης και αναλαμβάνει την αρμοδιότητα ε, να ερευνά τις υποθέσεις κάθε φορά που το κρατικό απόρριτο προβάλλει το εμπόδιο στην δικαστική εξουσία. Το κόπεσιτ αυτή αυτά τα χρόνια δεν έχει βρει ούτε μία φορά να έχει υπάρξει υπέρβαση του κρατικού απορρίτου και ούτε μπορεί να το ανακαλέσει, διότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες εδώ. Ο δικαστικός έλεγχος που αναλαμβάνει το ε, συνταγματικό δικαστήριο έχει να κάνει με το κατά πόσον μια δικαιοδοσία θεωρεί ότι υπάρχουν αποδείξεις για υποθέσεις όπου έχει επιβληθεί το κρατικό απόρριτο ότι εκεί αδικαιολόγητα έχει γίνει η επίκληση του κρατικού απορρίτου. Τότε μπορεί να υπάρξει ε, προσφυγή στο δικαστήριο αυτό εφόσον θεωρηθεί ότι κάτι συγκαλύπτεται από το κρατικό απόρριτο από την εκπληκτική εξουσία. Ε, κυρίε και κύριοι, στην Ιταλία το κρατικό απόρριτο στην υπόθεση Αμπού Ομάρ Το επικαλέστηκαν όλες οι κυβερνήσεις ε, από την πρώτη και μετά. Ε, Πρόντι, ε, Μπερλουσκόνη, Ενολέτα, ε, Ρέντσι και τώρα για μια παρόμοια υπόθεση, διότι Ήδη βρήκα ονόματα δημοσιογράφων, δικαστών, πολιτικών ε, στελεχών που σε κάποιες περιπτώσεις κατάχρησης κατέληξαν να εκδικάζονται από δικαστήρια της Περούντζα και εκεί ο Ρέντζ επικαλέστηκε το κρατικό απόρριτο. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ μιλάμε για συγκάλυψη πληροφοριών, υποκλοπών, ε, γράφων και με την μεγάλη αυτή υπέρβαση του αρχικού ορισμού του κρατικού απορρίτου και κάποιες φορές ε, οδηγούν και σε κομικοτραγικές καταστάσεις και το κρατικό απόρριτο το έχουν επικαλεστεί για κάποιες περιπτώσεις διαφθοράς, δωροδοκίας, ε, οργάνωσης εγκληματικής. Αυτά ε, δεν μπορεί να τα επικαλεστεί κανείς για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Επίσης, Δύο από τους πρώτους προέδρους της Επιτροπής ήταν και ε, μέλη του Υπαρχικού Συμβουλίου και εκεί ε, επικαλέστηκε πάλι το κρατικό απόρριτο πρώτη. Να προχωρήσω. Για την έκθεση της Επιτροπής και την έρευνα της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Νόμοι στην Ιταλία λοιπόν υπάρχουν. Μπορεί να είναι ωραιότατα σχεδιασμένοι, αλλά μετά δεν υπάρχει ο πολιτικός και ο δικαστικός έλεγχος που προβλεπόταν στην Ιταλία έχει συμβεί με την τελευταία αντιπαράθεση των κυβερνήσεων ε, Πρόντι και Λέτα, Μόντι και Λέτα, να μην ασκηθεί το κρατικό απόρριτο. Το ακυρωτικό δικαστήριο λοιπόν αναγκάστηκε να ολοκληρώσει τη δίκη με πολύ σκληρέ διατυπώσει κατά του συνταγματικού δικαστηρίου. Έχουμε λοιπόν μια ανοιχτή δρυμή αντιπαράθεση μεταξύ συνταγματικού και αδικαιωτικού δικαστηρίου. Η μελέτη που υποβλήθηκε προηγουμένω, που παρουσιάστηκε προηγουμένω, είναι κατά με εξαιρετική σημασία. Θα καλούσα το κοινοβούλιο να το μεταφράσει σε όλε τι ε, επίσημε γλώσσε και να το διαδώσει. Να τη διαδώσει, διότι πραγματικά έχει εξαιρετική σημασία. Έχει κάποιε ανακρίβειε για την υπόθεση Αμπουομάρ και είμαι πρόθυμο να στείλω γραπτά κάποιε διορθώσει, αλλά μου φαίνεται σημαντικό να ε, όλα αυτά που επιβεβαιώθηκαν για ιστορικού λόγου να καταγραφούν και να γίνουν γνωστά. Επίση, μιλούμε για χειραγώγηση των δικαστηριών. Άκουσα προηγουμένω από την κυρία Γκόμε τα λόγια τη για την κυρία Σόζα. Εδώ Εδώ λοιπόν είδαμε ότι στην Ιταλία ε, θα μπορούσαμε να έχουμε χειριστεί πολύ διαφορετικά τα πράγματα, τις ειδίκες αυτές, εάν είχαμε διαφορετική ε, ευθύνη για το βάρο της απόδειξης. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι να αφήνουμε τα μεγάλα ψάρια πιάνοντα τα μικρά όπω είπατε, αλλά να υπάρχει ισοτιμία ενώπιν τη δικαιοσύνη για όλους. Πάντως στην έκθεση ΛΥΜΠΕ σωστά υπογραμμίζεται η ε, έλλειψη της δικαστικής συνεργασίας το Ιταλικό Δικαστήριο δεν στέλνει εύκολα αιτήματα για δικαστική συνεργασία πέραν από τα αιτήματα για παραδόσεις. Πάντως η έκθεση Φάινστάιν ε, εντοπίζει και μία, ε, κάτι το περίεργο για, τις, ε, κρατικές, για τα κρατικά έγγραφα. Γιατί δεν αναφέρεται πουθενά η υπόθεση Αμπού Ομάρ. Το πρόβλημα δεν είναι, υπήρξαν, δεν είναι ότι υπήρξαν απλώς 26 αμερικανικές καταδίκες εκρεμεί και άλλο αίτημα χάριτος ε, ενώπιον του ε, Ανώτατου Δικαστηρίου και υπάρχουν και άλλα αίτηματα από αυτούς που έχουν καταδικαστεί. Το θέμα είναι ότι η έκθεση Φέινσταϊν δεν μιλά ούτε για τις Ιταλικές υπηρεσίες στην Ιταλία. Παρόλο που και η Ιταλία ερευνήθηκε. Να κλείσω εδώ την παρουσίασή μου. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πως η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ έχει, πολλα, προχωρήσει πολλά ψηφίσματα και μελέτες και σωστά καλεί να μελετηθούν. Θα συμφωνήσω με αυτά που είπαν ε, η κυρία Ίντφελ και ο κυρίος Κοέλιου, ότι δηλαδή έφτασε η στιγμή, και εδώ μιλώ ως πολίτης, να ζητήσουμε και κάτι διαφορετικό από το Κοινοβούλιο. Και το κάνω ε, με όλο το σοφασμό για το εξαιρετικό σας έργο και πραγματικά όσο το δυνατόν πιο ταπεινά, αλλά έχω μελετήσει τουλάχιστον 18 ψηφίσματα εκθέσεις μελέτες του Ευρωκοινοβουλίου και ε, στοιχεία έγγραφα από το Συμβούλιο της Ευρώπης που είναι δημοσιευμένα και στον ιστοτοπό του και υπάρχουν τουλάχιστον 34 μνήες παραπομπές σε τη δράση της, Επιτροπής, της έκτατης Επιτροπής του Κοινοβουλίου. Να θυμίσω και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εδώ και λίγο, ένα πολύ μικρό διάστημα έκλεισε η πρόσφατη υπόθεση, αλλά τουλάχιστον εδώ και 10 χρόνια, όπως είπατε, η Washington Post κατέγγειλε το γεγονός ότι η CIA είχε φυλακίσει και βασανίσει μέλη της υποτιθέμενης ε, έγιναν διάφορες έρευνες έκτοτε και πρέπει να πω ότι ήδη στην έκθεση της Επιτροπής, μάλλον η έκθεση Θάβα της ε, Βεροσονής Επιτροπής του Κοινοβουλίου, ε, αναφερόταν στο τέλος της σε έναν μηχανισμό, μηχανισμό που θα μπορούσε να, προφυ... να επικαλείται το άρθρο 7 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης. Ένα μηχανισμό δηλαδή προειδοποίησης για την περίπτωση κινδύνων ή κυρώσεων εφόσον δεν γίνονται σεβαστές οι θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης όπως προβλέπονται στο άρθρο 2. Και αυτό έχει συμπεριληφθεί στο ψήφισμα. Στο ψήφισμα που, που επαναλήφθηκε και από τον Δικ ε, Μάρτι εδώ λοιπόν με την ε, περιβόητη πλέον απόφαση Safe Harbor του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου βλέπουμε ότι το δικαίωμα αυτό ε, κάνει μια εκρηκτική εμφάνιση στο πολιτικό προσκήνιο. Όχι μόνο... Ε, όχι μόνο ως ε, συμβολική αξία, αλλά η, απόφαση του δικαστηρίου μας δείχνει ότι δεν μπορεί να παραγωνίζεται ο δικαστικό τομέας ε, και δικαστικές αποφάσεις ούτε στο όνομα οικονομικών συμφερόντων, ούτε εσωτερικών, ούτε υποτιθέμενης δημόσιας τάξης, φτάνει η αποσιώπηση των ε, βασανιστήριων, φτάνει η αποσιώπηση που επιβάλλει το κρατικό απόρριτο. Εδώ ουσιαστικά πρόκειται για απόπειρε συγκάλυψη από τι διάφορε κυβερνήσει και αυτό είναι μια πάγια πρακτική. Εδώ προσοχή, ε, μιλώ για την Ιταλία προφανώ, ένα λεπτό και τελειώνω πρόεδρε. Η Ιταλική κυβέρνηση, οι Ιταλικέ κυβερνήσει, ανέφερα πέντε, στην ε, υπόθεση Αμπου Ομάρ επεκαλέστηκαν το κρατικό απόρριτο επιβεβαίωσαν ε, προστρέχοντας το συνταγματικό δικαστήριο για να κλείσουν οι έρευνες μετά τις, τα δικά σας ψηφίσματα, μετά τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οπότε τι συμβαίνει. Απλές εξαγγελίες, ε, το Κοινοβούλιο υπήρξε, ανέλαβε το ρόλο της Κασάνδρας, υπήρξε πραγματικά διορατικό, είδε πολύ μακριά τον, στον ζωτό του χρόνου. Εάν είχε σταματήσει το Κοινοβούλιο και δεν πίεζε, όπω νομίζω θέλει να κάνει, την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναλάβουν τι αρμοδιότητε τους, και να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο και να γίνουν περαιτέρω βήματα, νομίζω ότι ως πολίτης μπορώ να πω ότι διακυβεύεται όχι μόνο η πρωτιά ενό θεσμικού οργάνου σε σχέση με ένα άλλο, αλλά και η πολιτική ισορροπία των διαφορών θεσμικών οργάνων μεταξύ του. Εμεί αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα Ευρωκοινοβούλιο που να μην είναι αδύναμο, όχι ότι είναι, αλλά ότι θα πρέπει να είναι ακόμα ισχυρότερο. Δεν μπορεί να προσπιστεί τα δικαιώματα των πολιτών που το ε, εξέλεξαν χωρί να φτάσει ω το τέρμα τη προσπάθειά του για να εξασφαλίσει την ισότητα. Η σύμβαση κατά των βασανιστήριων έχει αναφερθεί επανειλημμένω δεν είναι απλώς ένα κείμενο που θέλουμε να το κορνιζώσουμε και να το κρεμάσουμε στους τοίχους και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 11 Φεβρουαρίου 2015 λέει ότι θέλει να αναθέσει στον Πρόεδρό του να ε, αποστείλει το ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή και αυτό δεν το λέω μόνο γιατί το διαβάζω εδώ στο κείμενο αλλά γιατί καλό είναι να κινητοποιηθούν αυτοί οι μηχανισμοί. Χρειάζονται λοιπόν περισσότερα από απλές εξαγγελίες. Όποιος παροβίασε δικαιώματα θα πρέπει να έρθει αντιμέτωπος με τις ευθύνες του. Μιλάμε για θεμελιώδη δικαιώματα και θα πρέπει να τον στήσουμε στον τοίχο. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να ζητήσει το Κοινοβούλιο από το Συμβούλιο και την Ευρώπη και να φτάσω στο τέρμα τη προσπάθειά του. Και επιτρέψτε μου, γιατί μιλώ μόνο για όσα γνωρίζω καλά, ε, παρατηρώ ότι υπάρχει μια συνέπεια κάποιων ε, ευρωβουλευτών, αυτών που εδώ στην Ευρώπη προσυπογράφουν αυτέ τι σημαντικέ αρχέ, αλλά στα κράτη προελευσή του και στην Ιταλία κάποιε φορέ, ιδίω στην Ιταλία, τηρούν ε, σιωπή. με τον Κλάουντιο Φάβα, ο οποίο συμπεριφερόταν με με ένα συγκεκριμένο τρόπο ε, μάλλον είχε την ίδια συμπεριφορά και στη χώρα του την Ιταλία και στην Ευρώπη, στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό δεν συμβαίνει συχνά, δεν είναι χαρακτηριστικό τη Ιταλική συμπεριφορά. Και θα κλείσω με λίγα λόγια ενό μια ομιλία που χθε ο ε, κύριος Ματαρέλα εκφώνησε χθε σε μια συγκέντρωση Ιταλών βουλευτών του ε, Ιταλικού Κοινοβούλιο. Πρέπει να φροντίσουμε φωνή της Ευρώπης να έχει κύρος, να εκφράζει αξίες και όπως η δημοκρατία, η ειρήνη και η ισότητα ενώπιον του κράτου δικαίου. Αυτοί είναι οι λόγοι για του οποίου η Ήπειρο μα ε, φαίνεται ένα λιμένα ασφάλεια πολλέ φορέ ε, και γι' αυτό πολλέ φορέ κάποιοι χάνουν τη ζωή του προσπαθώντα να φτάσουν ακριβώ εδώ. Δεν αρκεί ω πρόσχημα η οικονομική κρίση ή το μεταναστευτικό κύμα ή οι απειλέ τη διεθνού τομοκρατία για να αλλάξει αυτό. Το είπε ο κ. Ματαρέλα. Νομίζω ότι ω ε, δικαστή ανακριτή μπορώ να το πω έχουν ακριστού και διάφορες ανοησίες βάσει του Μητρώου Επιβατών. Δεν χρησιμεύουν σε τίποτα, παραβιάζουν το αρνητικό βίο των πολιτών και το είπε και το ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ελπίζω λοιπόν εσείς να είστε εκείνοι που θα κρατήσετε ψηλά τη σημαία αυτή, να συνεχίσετε, να συνεχίσετε μπροστά ε, και να μην σταματήσετε. Και ε, να θυμίσω απλώς και τον Ισπανό συγγραφέα που τόσο πολύ μου αρέσει, τον ε, Σερκάς και να πω καλή τύχη. Ελπίζω να αναλάβετε ενεργό δράση για όλες αυτές τις ε, δράσεις που χρειάζονται ώστε τα ένοχα κράτη να, ε, αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και εφόσον χρειαστεί και τιμωρία, ας υπάρξει και τιμωρία, ας υπάρχουν κυρώσεις. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε αν ξέφυγα κατά τέσσερα λεπτά. Παρακαλώ. Ήταν ε, πολύ ωραία παρουσίασή σας με μεγάλο πάθος και ε, μιλήσατε για αυτό που σας ζητήσαμε, τη περίπτωση Αμπού Ομάρ αλλά μας είπατε και για την έκθεση ΦΑΒΑ, θέσατε το γενικότερο πλαίσιο, την ε, ε, ε, Εξεταστική Επιτροπή που προείδρευε ο κύριος Κοέγιο, θέσατε τη γενικότερη εικόνα και το γενικότερο πλαίσιο, το ιστορικό και πού βρισκόμαστε σήμερα και έχουμε εμείς τις ευθύνες. Και μας βοηθάει πάρα πολύ για τη σημερινή συνεδρίασή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα πρέπει να σα πω ότι δυστυχώ η καθηγήτρια κυρία Ντάφη ε, κολλεί τη τελευταία στιγμή ακύρωση την παρουσία τη και θα δώσω το λόγο στην τελευταία μα ομιλήτρια που είναι η κυρία Σίνγκ και είναι αρμόδια για την καταπολέμηση τη δημοκρατία ε, και ε, την εθνική ασφάλεια, ε, ασχολείται με θέματα στρατηγικής ασφάλειας, κατά πολέμης τροποκρατίας, ανθρώπινα δικαιώματα και βεβαίως συμπεριλαμβάνεται εδώ η παράνομη παράδοση, βασανιστήρια και κράτηση. Έχετε το λόγο και σας ευχαριστώ που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Είμαι ευγνώμων για τη δυνατότητα αυτή που μου δίνεται να μιλήσω εδώ σήμερα σε τούτη την ακρόαση. Η ακρόαση από μόνη της είναι ένα ε, γεγονός που επικροτούμε και ελπίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να πιέζει για λογοδοσία στις ε, ενέργειες της CIA όσον αφορά τις έκτακτες παραδόσεις ε, και τις μυστικές κρατήσεις. Έχω εργαστεί πάνω στο θέμα αυτό και από την πρόπτικη των ΗΠΑ και από την πρόπτικη της Ευρώπης ασχολούμαι με το θέμα αυτό από το 2001 και μετά και έχω συγγράψει και μία ε, έκθεση η οποία έχει να κάνει με την παγκοσμιοποίηση των βασανιστήριων, όπως είναι ο τίτλος της, ε, που έχει να κάνει με τον μεγάλο αριθμό κυβερνήσεων που συνεργάστηκαν σε αυτές ε, τις δραστηριότητες της CIA. Επιπλέον, ήμουνα δικηγόρος του κυρίου Αλνάσρη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην ε, υπόθεση κατά Πολωνίας, ε, την οποία κερδίσαμε. Ήταν πολύ μεγάλη σημασία αυτή η απόφαση της 24ης Ιουλίου του 2014. Και επίσης ε, τον εκπροσωπώ στην υπόθεση κατά της Ρουμανίας που εκκρεμεί ακόμα. Στο προηγούμενο πάνελ ακούσαμε ότι είναι σαφές ότι οι υποθέσεις αυτές κατά Πολωνίας και κατά Ρουμανίας αποτελούν μέρη του ιδίου πλαισίου και της ίδιας νομικής υποδομής όσον αφορά δηλαδή την ανάλυση των ενεργειών της CIA στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε δύο πολύ σημαντικές αποφάσεις του ε, ΔΕΚ. Η, μία, η πρώτη κατά το, της Μακεδονίας και η δεύτερη κατά της Πολωνίας ε, που και οι δύο εκδόθηκαν ε, την ίδια μέρα. και η Μακεδονία και η Πολωνία να θεωρούνται υπεύθυνε τις δύο χώρες αυτές υπεύθυνε για έκτακτες παραδόσεις και μυστικέ κρατήσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι οι ε, αποφάσεις επειδή απαγορεύουν τη συνεργασία ε, ευρωπαϊκών ε, κρατών σε αυτές τις καθαρά παράνομες ενέργειες, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσο θα συμμορφωθούν τα κράτη-μέλη με τις αποφάσεις. Απομένει δηλαδή ακόμα να δούμε αν η κυβέρνηση της Μακεδονίας και της Πολωνίας θα διεξάγουν ε, αποτελεσματικές έρευνες όπως ε, απαιτεί η απόφαση του δικαστηρίου. Και στην περίπτωση της ε, Μακεδονίας και στην περίπτωση της Πολωνίας το δικαστήριο απεφάνθη ότι οι κυβερνήσεις είχαν αποτύχει όσον αφορά την, σημαντική, την σωστή διερεύνηση των κατηγοριών. Υπάρχουν λοιπόν σημαντικά ε, ερωτήματα παρά τις αποφάσεις αυτές όσον αφορά την εφαρμογή τους, την εκτέλεση των αποφάσεων. Πιο πρόσφατα, τον Μάρτιο του 2015, ε, ε, η Υπουργή Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με τον ε, κύριο Ανάσο, διότι κρατείται αυτή τη στιγμή στο Κουαντάναμο υπάρχει απειλή ότι θα δικαστεί από, από τη Στρατιωτική Επιτροπή και ότι θα καταδικαστεί σε θάνατο. Θα ήθελα να επιθύσω την προσοχή σα στο γεγονό ότι αυτέ οι υποθέσει έκτακτων παραδόσεων και μυστικών κρατήσεων αφορούν όχι μόνο το άρθρο 2, συγγνώμη, άρθρο 3, διορθώνει ομιλήτρια της σύμβαση για τα Βασανιστήρια, αλλά και ε, το άρθρο 2 που έχει να κάνει με τη θανατική ποινή. Και στην υπόθεση Αλάσσοη κατά Πολωνίας, ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, είπε ότι είχε ε, παραβιαστεί το άρθρο 2 επειδή είχε βοηθήσει η Πολωνία την ε, μεταγωγή ε, του κυρίου Αλνασρή για να αντιμετωπίσει την θανατική ποινή. Το ίδιο θέμα εμφανίζεται στην υπόθεση κατά που εκκρεμεί. Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις όχι μόνο μυστικές μυστικής ε, κράτησης ε, και βασανιστήριων σε ε, ρουμανικό έδαφος, αλλά και η βοήθεια της ρουμανικής κυβέρνησης προς τις ΗΠΑ για την μεταγωγή του κυρίου Αλτασρή, τη μεταφορά του δηλαδή εκτός Ρουμανίας. Θα ήθελα λοιπόν το Κοινοβούλιο να δώσει πολύ προσοχή στι στις υποθέσεις αυτές, διότι αποτελούν πολύ σημαντικές παραβιάσεις της Ευρωπαϊκή Σύμβαση και του Διεθνούς Δικαίου. Όσον αφορά την έκθεση της Γερουσίας, όπως, ε, πολύ, ε, όπως επανειλημμένα τόνισε το προηγούμενο πάνελ, ε, είναι πέραν κάθε αμφιβολίας ότι υπήρχε κατάσταση μυστικών κρατήσεων στην Πολωνία, ότι υπήρχε επίσης τέτοια κατάσταση στη Ρουμανία και επίσης έχει ε, αποδειχθεί πέραν ε, καθελοκής αμφιβολίας ότι υπήρχε ε, τέτοια κατάσταση στη Λιθουανία και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί μόνο από δημοσιογράφους αλλά και από την σχετική έκθεση και από τον αρμόδιο τα ανθρώπινα δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μάλιστα υπήρχε χαρτοφυλάκιο το οποίο περιείχε ε, αποδεικτικά στοιχεία και ο κύριος Χάμερπερκ δεν έλαβε απάντηση στο σχετικό του αίτημα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό. να δούμε τις παρατηρήσεις της κυρίας Ευαζολή στο ευρύτερο πλαίσιο της πρακτικής της Ρουμανίας, της πρακτικής άρνησης της Ρουμανίας. Και ε, αυτό έχει τεκμηριωθεί στην, στα έγγραφα που έχουμε δώσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ήταν ε, συνεχής πρακτική της, ε, των Ρουμανικών αρχών να αρνούνται την ύπαρξη των μυστικών φυλακών. Και αυτό μας ενδιαφέρει αντικειμενικά, το ότι δηλαδή αρνούνται την ύπαρξη παρά τα σαφή αποδεικτικά στοιχεία. Και δεν είναι αξιόπιστη η στάση της Ρουμανίας. Αλλά η συνεχής αυτή άρνηση θέτει και το πλαίσιο εντός του οποίου η Ρουμανία επιδεικνύει έλλειψη βούλησης να διεξάγει αποτελεσματική έρευνα. Στην υπόθεση Αλνασρή κατά Πολωνία είχαμε ακριβώ αυτό. Σημασία έχει όχι μόνο αυτό που λέει σήμερα ή που θα πει αύριο η κυβέρνηση της Ρουμανίας, θα πρέπει να δούμε και την ε, πρακτική της κυβέρνησης στο παρελθόν. Και μάλιστα στο τελευταίο αυτό πάνελ, αλλά και στο προηγούμενο έχει αναφερθεί επανειλημμένα το γεγονός ότι το 2005 η Human Rights Watch διαπίστωσε ότι υπάρχει εγκατάσταση για μυστικές κρατήσεις στη Ρουμανία. Εάν εξετάσουμε την πρακτική άρνηση της ρουμανικής κυβέρνησης έκτοτε, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει καμία βούληση να διεξαχθούν αποτελεσματικές έρευνες. Στην υπόθεση λοιπόν Αλνασρή κατά Πολωνίας, ε, βγάζουμε το ε, συμπέρασμα ότι η Ρουμανία έχει ε, καταστρατηγεί στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση όπως και η Πολωνία. Αυτό είναι λογικό συμπέρασμα. Καλό λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να το σημειώσει αυτό. Τα γεγονότα σε σχέση με τη Ρουμανία ε, αποδείχθηκαν όχι μόνο με την έκθεση της ε, Γερουσίας, αλλά όπως είπε και ο κύριος Μπλακ πριν την δημοσίευση της έκθεσης αυτής, διότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο άκουσε τις μαρτυρίες του Γερουσιαστή Μάρτη και ενός εμπειρογνώμονα που επιβεβαίωσαν ότι υπήρχε φυλακή στη Ρουμανία και η απόφαση αυτή ήταν του Ιουλίου του 2014 πριν δηλαδή την ε, δημοσίευση της ε, έκθεσης της Γερουσίας. Η έκθεση της Γερουσίας επιβεβαιώνει ότι από το 2003 ε, μέχρι, το 2000, μέχρι τον Νοέμβριο του 2005 λειτουργούσε η εγκατάσταση αυτή στη Ρουμανία και το δικαστήριο θεώρησε ότι είναι αδιανόητο η Ρουμανία να έχει... Η Ρουμανία να έχει μια τέτοια... Η Πολωνία να έχει μια τέτοια εγκατάσταση ε, χωρίς την γνώση των ε, αρχών, έτσι είναι αδιανόητο και στη Ρουμανία αυτό και η έκθεση της Γερουσίας παρουσιάζει σαφή αποδεικτικά στοιχεία ε, που στηρίζουν το συμπέρασμα αυτό. Δείχνουν ότι οι χώρες αυτές ήρθαν, ε, ε, συνήψαν συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την δημιουργία τέτοιων εγκαταστάσεων και ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε πλήρωσαν πάνω από 8 εκατομμύρια δολάρια στις αρχές της Ρουμανίας. Εάν λοιπόν η Ρουμανία δεν γνώριζε τίποτα γι' αυτό, πώς είναι δυνατόν η έκθεση της Γερουσίας να αναφέρεται σε συμφωνία, να αναφέρει εκατομμύρια δολάρια που δόθηκαν στις αρχές της Ρουμανίας. Έτσι τίθενται πολύ σοβαρά ερωτήματα σχετικά με αυτές τις έρευνες στη Ρουμανία. Θα ήθελα να προσθέσω ότι ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απαιτεί η έρευνα να είναι ποινική φύση για να ε, εξεταστεί υπό το άρθρο 3 της ε, σύμβασης και οι έρευνες αυτές δεν ξεκίνησαν παρά μόνο μετά την ποινική δίωξη που άσκησε ο κύριος Αλνασρή το 2008 και είναι πάρα πολύ σαφές ότι τα κράτη έχουν υποχρέωση από μόνα τους ε, να διεξάγουν έρευνα τη στιγμή που ε, προκύπτει μια τέτοια υπόθεση και ξέρουμε ότι το Νοέμβριο του 2005 υπήρχε τέτοια υπόθεση. Μάλιστα οι αρχές της Ρουμανίας πριν το 2005 ε, γνώριζαν ότι είχαν στο έδαφος τους μυστική φυλακή, διότι ε, υπήρχε η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβετε ότι υπήρχαν παράγοντες εντό στις ρουμανική κυβέρνηση που γνώριζαν ότι έχουν συμβεί αυτό. Είναι αδιανόητο να μην το γνώριζαν. So I would just end θα ήθελα λοιπόν να κλείσω τονίζοντας αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές, ότι υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι υπήρχαν τέτοιες μυθείς καταστάσεις στην Πολωνία, τη Ρουμανία και την Λιθουανία και ότι πολλά κράτη-μέλη συνεργάστηκαν με την CIA είτε επιτρέποντας υπερτήσεις ε, είτε με άλλους τρόπους και είναι πάρα πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεχίσει να, να ασχολείται με το θέμα, να λάβει την ε, εντολή και τους, το δυναμικό που απαιτείται ε, για να απαιτήσει λογοδοσία σε αυτήν την πολύ σημαντική παραβίαση του κράτους δικαίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα αρχίζει η συζήτηση. Ο κύριος Κορέγιο πρώτος. Ευχαριστώ. Queria agradecer ao juiz Patário e à Singh as intervenções. Ευχαριστούμε για τις ομιλίες σας και κυρίως τον κύριο Σπατάρο. Ξέρει ότι, είναι, ότι είμαι θαυμαστής του, της δουλειάς του. και η ανάκριση που έφερε πέρας έκανε πραγματικά τη διαφορά στο πώς ε, φαίνεται η εικόνα της Ευρώπης. Διότι πολλοί από εμά ε, φράζουμε τη λύπη μας για την έρευνα κοινοβουλευτικών έρευνων και δικαστικών έρευνων και δικαιολογημένα και το γεγονός ότι υπήρξε μια ε, ολοκληρωμένη δικαστική έρευνα από τον ε, δικαστή Σπατάρο δείχνει ότι η ατιμορρησία δεν είναι πάντοτε κανόνας αυτή που ίσχυσε σε πολλές περιπτώσεις. Όποιος λοιπόν ε, παραβιάζει τον νόμο και τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορεί να τιμωρείται και χαίρομαι ιδιαίτερα για τον ενθουσιασμό με τον οποίο υπερασπίστηκε την δικαστική έρευνα ο δικαστής Σπατάρο και με την εξουσία και το κύρος που έχει μας θύμισε ότι ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Εδώ λοιπόν δεν πρόκειται να σταματήσουμε να διαδραματίζουμε το ρόλο μα, ιδίω εγώ ίδιο όσο μπορώ να δεσμευτώ με κάθε συνέπεια. Απλώ υπάρχουν μερικά θέματα που ξεφεύγουν των δικών μα αρμοδιοτήτων. Σωστά είπε ο κ. Πατάρο ότι υπάρχει κατάχρηση του κρατικού απορρίτου. Ότι οι μηχανισμοί ε, εθνικού ελέγχου, οι εθνικοί μάλλον μηχανισμοί ελέγχου, για το κατά πόσον υπάρχει ε, παραβίαση ή όχι, στι περισσότερε περιπτώσει δεν χρησιμοποιούνται σωστά. Να προσθέσω και το εξή Κάτι που το έχουμε ε, εξετάσει επανειλημμένως και που ήδη έχει απασχολήσει την Επιτροπή μας. Δεν υπάρχει ε, ε, συνεκτικότητα, συνοχή στον έλεγχο των μηχανισμών αυτών του κράτους. Είτε στο δικαστικό, από την πλευρά του δικαστικού, είτε του κυβερνητικού ελέγχου. Οι κανόνε βέβαια είναι πολύ διαφορετικοί μεταξύ των χωρών. Σε κάποιε χώρε δεν υπάρχει κανένα είδου έλεγχος, κάποιοι έχουν και τα δύο είδη, κάποιοι έχουν ψεύδο ελέγχου κάποιοι που μπορεί να καλύπτονται από, ή να προβλέπονται από τον νόμο και μετά τελικά στην πράξη να μην γίνονται ποτέ πραγματικότητα. Όμως δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι νόμοι των κρατών μελών πολύ συγκεκριμένα. Μάλλον δεν έχουμε κανένα λόγο συγκεκριμένα στον έλεγχο για το κρατικό απόρριτο μπορούν να κάνουν τα εθνικά κράτη. Είναι εθνική αρμοδιότητα αυτή. Τα εθνικά κράτη με τους εθνικούς τους βουλευτές επιτρέπουν απλώς να υπάρξει μια ανταλλαγή απόψεων, διάλογος και έτσι έχουν δημοσιευθεί και κάποια έγγραφα του Κοινοβουλίου σε σχέση με το θέμα αυτό. Πέραν αυτού όμως και όσο και αν θέλαμε να πάμε πέρα από τις αρμόδιότητές μας και όσο και αν υπερασπίζεται με ενθουσιασμό δικαστής Πατάρο τον άμεσο έλεγχο και εργάζεται στο πλαίσιο όσων προβλέπει ο νόμο, ε, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορείτε κι εσεί να μα ζητήσετε να υπερβούμε δυστυχώ τι αρμοδιότητέ μα και να αναλάβουμε πράγματα για τα οποία δεν έχουμε καμία εξουσία. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Γκόμες Και εγώ θαυμάζω πάρα πολύ το έργο του δικαστού Σπατάρο στην Ιταλία και βεβαίως για μας ήταν ουσιαστικό για να καταλάβουμε τι διακυβεύεται. Και είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στον κύριο Σπατάρο, διότι ήρθε εδώ ακριβώ να μας πει αυτό, ότι η κατάχρηση του κρατικού απορρίτου είναι κάτι που αποτρέπει τους υπευθύνου να λογοδοτούν. Το είπε και ο Κάρλος Κόγια, ότι δεν είναι δική μας δουλειά να αποφασίσουμε για το πώς χρησιμοποιεί και επικαλείται το κρατικό πόρη κάθε χώρα. Αλλά δουλειά μας είναι να πούμε στις κυβερνήσεις μας ότι κάνουν κατάχρηση του κρατικού απορρίτου και των κρατικών μυστικών ακριβώς για να εμποδίσουν τη διερεύνηση και για να συγκαλύψουν εκείνους τους πολιτικούς σε υψηλούς τόκους που ευθύνονται και επικεφαλής μυστικών υπηρεσιών και υπαλλήλου μυστικών υπηρεσιών που είχαν διαταγές να ε, συμμετέχουν και να συγκαλύπτουν αυτά τα προγράμματα κράτησης και βασανιστήριων. Και αυτό θα πρέπει να βγει ως συμπέρασμα και να είναι συνέπεια της δικής μας ακρόασης σήμερα. Δεν συμβαίνει μόνο στην Ιταλία, σε άλλες χώρες και στη Ρουμανία, ο Κάλλος Κόγιο και εγώ ήμασταν μέλη της πρώτης αντιπροσωπείας που μετέβη το 2007 στη Ρουμανία και γυρίσαμε πίσω απολύτως πεπισμένοι ότι ε, το γνώριζαν οι Ρουμάνοι. Ορισμένοι μας είπαν και αντιφατικά πράγματα. Βρήκαμε ένα ε, υπάλληλο μυστικών υπηρεσιών και τελικά μας είπε ότι υπήρχαν διάφορες μυστήριες διαδρομές πτήσεων και τα λοιπά και στην ε, Κωνσταντσα ας πούμε κοντά υπήρχε μια μυστική φυλακή. Δηλαδή, οι Ρουμάνοι συνάδελφοι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ε, και του δικού μου, σας λέω σταματήστε να αρνείστε ότι συνέβησαν αυτά, μα τα γνωρίζουμε ότι έχουν γίνει. Αναλάβετε τις ευθύνε σας επιτέλους και να βρούμε αυτού που είναι οι υπεύθυνοι. Και επανέρχομαι στη δική μου χώρα, την Πορτογαλία, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, προσέξτε το. Το είπε και η καθηγήτρια mm. Γκίλτ προηγουμένως. Για ποιο τρόπο και με ποιο τρόπο στην Πολωνία επελέγει η συγκεκριμένη μυστική υπηρεσία που ήταν του στρατού. Η CIA δηλαδή επέλεξε τις στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες και πληροφοριών. Και στην Πορτογαλία δεν είναι μόνο μυστικές υπηρεσίες, είναι και οι ενοπλές δυνάμεις. Και το λέει αυτό και η έκθεση ΦΑΒΑ υπάρχει αναφορά για τον κατάλογο πτήσεων που πέρασαν από πορτοκαλικούς αερολιμένες με τη συνενοχή των στρατιωτικών και δεν ήταν μόνο πολιτικές πτήσεις, ήταν και στρατιωτικές πτήσεις. Της πολεμικής αεροπορίας δηλαδή δεν ήταν ε, ε, η συνενοχή μόνο των μυστικών υπηρεσιών έτσι και αλλιώς αλλά και των στρατιωτικών. Αυτό είναι πάρα πολύ βαρύ και σοβαρό. και στην χώρα μου ήταν κυβέρνηση δική μου ε, τότε και με κατηγόρησαν ότι ήμουν ψεύτρα καθόλου εκείνοι απεδείχθησαν ψεύτες είναι πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να τα αγνοούμε ή να υποκρινόμαστε ότι δεν τρέχει τίποτα υπάρχουν ευθύνε υψηλά εισαμένων προσώπων και θα πρέπει να αποδοθούν ευχαριστώ Αυξήθηκε ο κατάλογος των ομιλητών στο μεταξύ. Λοιπόν, σχολάρε και διερμηνείς κάποια στιγμή, έτσι, παρακαλώ το έχουμε υπόψη μας αυτό. Η κυρία Κουντρίτσκα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι δεν χωρά καμιά αμφιβολία ότι το 2002 και το 2003 οι πολωνικές υπηρεσίες προφοριών ναι. συνεργαζόντουσαν με την CIA σε ό,τι αφορά τα κέντρα αυτά κράτησης. Το πρόβλημα ποιο είναι όμως. Το πρόβλημα είναι ότι τα βλέπουμε όλα αυτά και τα εξετάζουμε πάρα πολύ επιπόλαια λέμε ότι η κυβέρνηση μπορούσε πραγματικά να παρέμβει, να συγκαλύψει, να καλύψει τους ε, υπεύθυνου και την αλήθεια. Ας θυμηθούμε ότι το 2008 στην Πολωνία εισήχθη η ανεξαρτησία του Γενικού Ισαντιλέα. Ε, γιατί στο παρελθόν υπαγόταν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Δηλαδή ο Γενικό Εισαγγελέα ήταν ε, ταυτόχρονα και Υπουργό Δικαιοσύνη, ήταν το ίδιο πρόσωπο. Τώρα έχει διαχωριστεί αυτό, υπάρχει διάκριση των εξουσιών και ε, η νυν κυβέρνηση επικρίνει πάρα πολύ τον Γενικό Εισαγγελέα. Λοιπόν, βλέπουμε ε, ότι η δυνατότητα επέμβασης των πολιτικών στη δικαιοσύνη είναι πάρα πολύ περιορισμένη και είναι καλό αυτό. Έχω λοιπόν δύο ερωτήσεις προς τον κύριο Σπατάρο. Είναι καλό αυτό ο εισαγγελέα και η εισαγγελία να είναι απολύτω ανεξάρτητη αρχή από την πολιτική ή όχι. Ακριβώ αυτή η διάκριση των εξουσιών εξασφαλίζει ότι δεν επεμβαίνει στην ε, δικαιοσύνη η εκάστοτε κυβέρνηση. Έχω και μια ερώτηση προς την κυρία Σινγκ. Εξ όσων γνωρίζω, η Πολωνία συμμορφώθηκε με την απόφαση ε, του ΕΔΑΤ. Στην αρχή κάναμε προσφυγή. Ε, στη συνέχεια καταβάλαμε την οικονομική αποζημίωση που ήταν 100.000 ευρώ αν δεν απατώμε. Αλλά εσείς γνωρίζετε αν κατέβαλε αυτό το ποσό η Πολωνία ή όχι. Την αποζημίωση. Εσείς που είστε και συνήγορος του κυρίου αυτού θα πρέπει να το γνωρίζετε. Αυτή τη στιγμή στην Πολωνία ε, ε, γίνεται αυτή η έρευνα την οποία ξεκίνησε ο κύριος Αλνάσρη ε, και είναι ακόμα καθοδόν και σύμφωνα με τη διάκριση των εξουσιών κατά Μοντεσκέ είναι απολύτως ανεξάρτητη η δικαστική εξουσία. Στην Πολωνία εμείς έχουμε να κατηγορήσουμε τη δικαιοσύνη για διάφορα, για χρονοτριβές, για πολύ μακροσκελείς διαδικασίες, αλλά Τώρα αυτή η υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη, δεν αναμειγνύεται η πολιτική. Είναι στα χέρια της δικαστικής εξουσίας και εκείνοι ε, θα τα διευκρινίσουν όλα αυτά τα πράγματα και θα διαλευκάνουν την κατάσταση. Εμείς ως πολιτικοί δεν μπορούμε να επέμβουμε. Γιατί αυτό θα ήταν πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό ως επέμβαση και στην εξαρτησία των δικαστήριων. Ευχαριστώ πολύ. Ο Φόιχτ. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση προς τον κύριο Σπατάρο. Είπατε ότι υπάρχει ήδη ε, μια αίτηση χάριτος ε, που έχει υποβληθεί ε, από έναν των 26 της CIA. Ποια χάρη για κάποιον βασανιστή και κάποιον που απαγάγει ανθρώπους και με εκπλήσει που 26 ε, αυτοί οι οποίοι είναι Αμερικανοί πολίτες ε, καταφέρατε να τους καταδικάσετε στην Ιταλία. Γιατί σήμερα το πρωί ε, επαναλάβαμε και ακούσαμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι υπέρ της ασυλίας όλων αυτών που συμμετείχαν σε απαγωγές και σε βασανιστήρια. Πώς καταφέρατε εσείς να τους καταδικάσετε στην Ιταλία. Ε, ήταν παρόντες ε, οι ίδιοι, ε, είχαν συνήγορο, υπήρχε δυνατότητα προσφυγής στο εφετείο, καταθέσαν έθεση έθεση Ευχαριστώ η κυρία Ινετσφέλτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε πολύ σύντομα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Σπατάρο για τη δουλειά του τόσα χρόνια. Το ίδιο και στην κυρία Σιν για τη δική της προσπάθεια. Πρώτη ερώτηση προς τον κύριο Σπατάρο. Ξεκινήσαμε με ένα αίτημα για παράδοση, για έκδοση από τις αρχές της CIA. Σε περιπτώσεις ατόμων θα μπορούσαν και να ε, είχαν απελευθερωθεί. Αυτό είναι περίεργο και αυτό που κυρίως με παραξενεύει είναι ότι οι χώρες της Ένωσης φαίνεται να είναι όλο και πιο πρόθυμες να εκδώσουν πρόσωπα προς τις ΗΠΑ παρά το αντίστροφο. Δεν θα έπρεπε να το δούμε αυτό και από την πλευρά των δικαστών. Μια προσφάτη υπόθεση στις κάτω χώρες έχει για πρώτη φορά έναν δικαστή που έχει φέρει έναν δικαστή να αρνηθεί την έκδοση ενός νεαρού που οι Ηνωμένε Πολιτείες υποπτεύονταν ότι ο που λέγανε ότι οι τουριστικές του δραστηριότητες ήταν ε, ύποπτες ε, και δεν εκδόθηκε γιατί δεν θα τύχει δίκης δίκης ε, και μπορεί να έρθει αντιμέτωπος και με τη θανατική καταδίκη λέει ο δικός μας δικαστή έτσι λοιπόν, γιατί οι εκδόσεις προς τις ΗΠΑ και όχι αντιστρόφως υπάρχουν δικαστές στις ΗΠΑ που να έχουν επικαλέσει το ίδιο και έπειτα να επαναλάβω την έκκληση της Άννας Γκόμες προς εμάς τους ιδίους κατά κύριο λόγο, γιατί καλό θα ήταν να τα κάνουμε πράξη αυτά που αγγελιζόμαστε ως κοινοβούλιο. Υπάρχουν πολλά ψηφίσματα από το Κοινοβούλιο για τα ζητήματα που συζητούμε και νομίζω ότι οι ομάδες που βλέπω γύρω μου δεν θα ψηφίσουν ανάλογα με τα όσα δηλώνονται εδώ. Εάν δούμε και την παρελθούσα νομοθεσία, αυτά που ε, έχουν ψηφιστεί και εγκριθεί δεν συνάδουν με αυτά που υπόθεκαν σήμερα εδώ. Καλό θα ήταν λοιπόν να δείξουμε συνέπεια με τα όσα λέμε, με τις αρχές και τις αξίες μας και να εγκρίνουμε μόνο νομοθεσία που να μπορεί να περάσει το τεστ της νομιμότητας και της συνταγματικότητας. Ιδάλλως, θα συνεχίσουμε αυτή την πολιτική ρητορία και θα πηγαίνουμε σπίτι μας πολύ ευχαριστημένοι με τους εαυτούς μας, αλλά η νομοθεσία μας, αυτή που θα περνάει, δεν θα συμφωνεί με όσα λέμε. Όταν λοιπόν ψηφίσουμε σήμερα το απόγευμα, ίσως όλοι καλό θα ήταν να εξετάσουμε ε, αμήλικτα τη συνείδησή μα και να ψηφίσουμε αναλόγω με το όσα μας επιτάσσει η φωνή τη. Ευχαριστούμε κύριο Σόγκορ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λυπούμε που δεν παρακολούθησα ολόκληρη τη συζήτηση, αλλά έπρεπε να πάω στην Επιτροπή Απασχόληση. Μια ε, ίσως ε, απάντηση στην ε, κυρία Γκόμεφ. Ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών στη Ρουμανία το 2003, ο κ. Τάπες, και σύμβουλος του Προέδρου, ε, παραδέχτηκε στη Γερουσία το 2014, ναι, και προσπάθησαν να τα στελέχη να το ε, αρνηθούν ότι υπήρξε προσωρινή κράτηση λοιπόν και εξήγησε λίγο τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτό συνέβη πριν μπούμε στο ΝΑΤΟ. Οπότε η Ρουμανία βελτίωσε λίγο τη συμπεριφορά της ε, στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων πριν ε, μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα σύντομο σχόλιο, αν επιτρέπετε τώρα. Μέχρι το 2003 ε, αγωνιστήκαμε για να πείσουμε τον τότε πρόεδρο ότι το ολοκαύτωμα υπήρχε και η Ρουμανία συμμετείχε διότι ως το 2003 το αρνείτο, το αρνείτο και αυτό. Και τελευταία λεπτομέρεια για το ζήτημα των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Ρουμανία παραμένει μη προτεραιότητα στη χώρα μου από την δική μου εμπειρία και επειδή είμαι μελό εθνοτικής μειονότητας εκεί, μπορώ να το πω πέραν πάση αμφιβολία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και από τα μέλη της Επιτροπής, ο κ. Λόπε Αγγιλάρ. Ε, ευχαριστώ. Μία δήλωση για το τι αισθήματο μου προκαλεί όλο αυτό το ζήτημα, αλλά και προσπαθώντα να διερευνήσω λίγο καλύτερα τα όσα μας ανέπτυξαν οι υποστηκλημένοι μας. Υπάρχει ένα περιορισμένο φάσμα ε, δικαστικών υποθέσεων. Είπατε, κύριε Σπατάρο, την άποψή για τον κοινοβουλευτικό και το δικαστικό έλεγχο. Βεβαίω, αυτό είναι και η ουσία του κράτους δικαίου. Όμως, ο αριθμός υποθέσεων που έχουν βραχθεί, ε, που έχουν εκδικαστεί από τη δικαιοσύνη το τι έγινε στην πράξη με αυτές τις παράνομες απαγωγές κρατήσεις και τις ε, ε λανθασμένες, τις παράνομες πρακτικές της CIA με τη συνεργασία των κατομελών είναι πολύ περισμένος αριθμός των ε, υποθέσεων. Και παρόλο που εδώ προσπαθήσαμε να προκαλέσουμε, να ταράξουμε τα νερά στο Κοινοβούλιο και παρά την κάθε μας προσπάθεια πρέπει να αποδεχτούμε ότι οι αντιδράσεις της κοινή γνώμης στα, στα διάφορα κατημέλη ήταν πολύ χλιαρές. Τι θα είχατε να πείτε λοιπόν για τον περιορισμένο αριθμό υποθέσεων που έφτασαν στη δικαιοσύνη και ως προς την ποιότητα της απόκρισης. Κατά την, κατά την αίσθηση μου η Ιταλική υπόθεση είναι αρκετά ε, σημαντική. Όμως ήθελα ε, τη δική σας την ε, εντύπωση για τις διάφορες δικαστικές υποθέσεις ως τώρα και για τον τρόπο με τον οποίο ελέγχθησαν κύριε Σπατάρο. Σας ευχαριστώ κύριε Σπατάρο, κυρία Σιν. Θέλετε να απαντήσετε, αλλά αν μπορείτε σε ένα πεντάλεπτο καθένας. Βέβαια μπορείτε να υπερβείτε το χρόνο αυτό, αλλά Πολύ λίγο αν γίνεται. Ε, αν θέλετε λοιπόν να προσπαθήσετε να απαντήσετε στις ερωτήσεις και να κάνετε και σχόλια για όσα ακούσατε. Ελπίζω να μην είναι τελείως ε, χωρίς καμία σειρά η απάντησή μου το τι είναι πιο δίκαιο ή όχι. Αν πρέπει ο εισαγγελέα δηλαδή να είναι τελείω ανεξάρτητο από την εκτελεστική εξουσία. Απάντηση για μένα είναι ναι. Χωρί εάν, χωρί μα και αλλά, χωρί καμία επιφύλαξη. Αυτό το θέμα όμω διαρκώ συζητιέται στην Ιταλία. Δεν έχει καμία σημασία από ποιο πολιτικό, ποια πολιτική πτέρυγα είναι η κυβέρνηση, από το κέντρο τα αριστερά και τα δεξιά. Όμω, Υπάρχει μια τάση να μην γίνεται αποδεκτό ότι μπορεί να είναι δικαστική εξουσία ανεξάρτητη. Στο καιρού του Μουσολίνη, το 1942 ο Ντούτσε μπήκε στην αίθουσα όπου ε, αναλάμβαναν καθήκοντα οι ανώτατε δικαστές και τον χαιρέτησαν με υψωμένο χέρι οι τότε αξιωματούχοι. Ο Ντούτσε είπε τότε ότι κάποιοι πολιτικοί λόγοι μερικές φορές πριτανεύουν, ε, περισχύουν εναντί της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας. Το είπα συνοψίζοντας. Τέλος πάντων στην Ιταλία κάποιοι πιστεύουν ότι η δικαστική εξουσία, τη διαφθορά, τις απάτες, όλες τις άλλες υποθέσεις πρέπει να τα λαμβάνουν και να τα εξετάζουν να τα λαμβάνουν υπόψη και να τα εξετάζουν βάσει των ε, όσων συμβαίνουν στην οικονομία μα. Λε και οι οικονομικέ επιταγέ μπορούν να καθορίζουν τι δικαστικέ έρευνε. Κι όμω το σύστημά μα προβλέπει δύο σημαντικότατα ποινά. Το πρώτο είναι ότι το Υπουργείο Εσωτερικών στην Ιταλία η εισαγγελία μπορεί να είναι τελείως ανεξάρτητη. Ο Υπουργός δεν μπορεί να μας δώσει καμία ένδειξη. Δεν το λέω αυτό ως φανατικός της ανεξαρτησίας μας, αλλά τουλάχιστον οι εγγυήσει της νομοθεσίας είναι εγγυήσει προς τους πολίτες, εγγυήσει ισότητας. Έπειτα, η οποιαδήποτε ποινική, η οποιαδήποτε ποινική ε, δίωξη στην Ιταλία δεν είναι προαιρετική, είναι υποχρεωτική. Δεν μπορώ λοιπόν για μια υπόθεση να διεξάγω έρευνα σε μια άλλη, όχι, για λόγους ε, σκοπιμότητας ή οποιοδήποτε άλλου λόγου. Ε, τρίτη παρατήρηση, το σύστημα προβλέπει η αστυνομία που κάνει την έρευνα, η αστυνομική αρχή, να εξαρτάται μόνο από εμά, όχι από το Υπουργείο Εσωτερικών, από το Υπουργείο Άμυνα, αλλά από την δικαστική εξουσία. Άρα να είναι και αυτή την ανεξάρτητη. Αυτό είναι το σύστημά μας. Η ανεξαρτησία λοιπόν δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. απαιτεί και τον ανάλογο επαγγελματισμό. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει και ανάλογη ετοιμασία και ε, εξειδίκευση. Γι' αυτό και το ακυρωτικό δικαστήριο μπόρεσε να εκφράσει μία κριτική κατά του συνταγματικού δικαστηρίου ότι πρέπει να εκριζωθεί τελείως η δυνατότητα να επικαλείται κανείς για ε, λόγους γιατί λογικοφανεί το κρατικό απόρριτο. Μία τοποθέτηση πολιτικού χαρακτήρα πολύ σημαντική. Και έγιναν και πολλές παρατηρήσεις από τον ε, κύριο Κοέλιου για την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, τη δυνατότητα ε, να παρέμβουν σε όλα αυτά οι βουλευτές και το πόσο περιορισμένες μπορεί να είναι οι του Ευρωκοινοβουλίου. Τα είπα ως ε, πολίτης, δεν τα γνωρίζω τα της πολιτικής επακριβώς, αλλά οι έξι συστάσεις με τις οποίες κλείνει η έκθεση που σχολιάσαμε, σε κάποιο σημείο τουλάχιστον, και μιλώ για τη δεύτερη σύσταση, μιλά για την ενεργοποίηση της διαδικασίας του άρθρου 7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει είτε την περίπτωση σοβαρής παραβίασης των αρχών ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από ένα μέλος Ε, οπότε το ίδιο το σύστημα, το εσωτερικό σύστημα του Κοινοβουλίου επιτρέπει να ενεργοποιηθούν αυτές οι διαδικασίες που προϋποθέτουν βέβαια την ε, δυνατότητα την ε, ερευνητική και ανακριτική του Κοινοβουλίου. Πρέπει δηλαδή να ερευνηθεί ακόμη και η πιθανότητα, ο κίνδυνος παραβίασης των ε, δικαιωμάτων αυτών. Θα μπορούσε λοιπόν να είναι λίγο πιο αποφασιστική η δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, δεν ξέρω αν θα είναι με νομοθετική δράση με ποιο τρόπο, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα να το πω αυτό, αλλά έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν δυνατότητες δράσης για το Κοινοβουλίο και μάλιστα σημαντικές. Ως προς την χάρη. 5 Απριλίου 2013 ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Τζόντον Απολετάνο, ε, προέβλεψε, ε, δέχτηκε το αίτημα χάριτος του, του Τζόζεφ Εδώ ε, υπήρχε η υποψία ότι το αεροδρόμιο του Αβιάνο διατέθηκε στις Αμερικανικές Αρχές για την απαγωγή του ε, Μπου. Αυτή ήταν η ανάμεξη στην υπόθεση αυτή. Ε, το δικαστήριο του Μιλάνου είχε τοποθετηθεί αρνητικά. Είχε γίνει αναφορά στις πρακτικές που θεωρήθηκαν παράνομες από την Ιταλία και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της ιστορικής αυτής της στιγμής όπου προέκυψε η τελική καταδίκη, Έχουμε να κάνουμε με ένα γεγονό που έχει και ιστορική σημασία. Υπάρχουν και νομικέ λεπτομέρειε τι οποίε δεν θα αναπτύξω γιατί θα είναι ιδιαίτερα περίπλοκε. Όμω Συνολικά η απόφαση αυτή προκάλεσε πολλά επικρατικά σχόλια, όχι μόνο από τους δικαστές αλλά και από τους νομικούς. Διότι τέλο πάντων αυτό που τελικώς αποφασίζει είναι, αυτός που τελικώς αποφασίζει είναι ο αρχηγός του κράτους. Και σίγουρα Υπάρχουν κι άλλες καταδίκες, όμως εδώ η Γενική Εισαγγελία δίνει την άποψή της. Ε, όχι οι δικαστές. Και βεβαίως τελικώς αποφασίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν στην ερώτησή σας αναφερθήκατε και στο πώς λειτουργεί όλη η διαδικασία ε, στην Ιταλία. Μπορείτε να τη διευκρινίσετε την ερώτησή σας για την ε, διαδικασία. Για τη δίκη ρώτησα, ε, είναι Αμερικανοί πολίτες αυτοί ε, τη CIA. Πώς, πώς μπορούν να καταδικάζονται. Είναι απόντες, ερήμην, καταδικάζονται, είναι παρόντες, έχουν νομική συνδρομή, συνήγορο, αυτό ρωτάω. Τέλεια. Πρόκειται για μια ερώτηση σημαντική. Διότι προηγουμένως είπα ότι η διπλωματική ασυλία δεν αναγνωρίστηκε σε πέντε διπλωμάτες ότι ασκούσαν δηλαδή τα διπλωματικά τους καθήκοντα για την ε, εκδίκαση ερήμην. Εδώ, εάν υπάρχει απόδειξη ότι ο Απόντας γνώριζε ότι εκδικάζεται η υπόθεση και υπάρξει και συνηγορός, μπορεί να γίνει εκδίκαση ερήμην. Αυτό συνέβη διότι κάποιοι είχαν διαφύγει ε, και ήταν ε, απόντες επειδή το επέλεξαν, όχι επειδή δεν γνώριζαν. Και υπήρξε και συνήγορο, ε, δικηγόρο που του περασπίστηκε δηλαδή και που κάποιε φορέ τον είχαν προσλάβει οι ίδιοι. Η κυρία Ιντβελτ ρώτησε για τι ε, εκδόσει. Να πω ότι εδώ ζητήσαμε από το Υπουργείο και 26 να εκδοθούν ή μάλλον να μεταφερθούν οι έρευνε, αλλά το Υπουργείο βάσει του συστήματό μα μπορεί να αρνηθεί το αίτημα αυτό. Αιτιολογήθηκε λέγοντας ότι μόλις το 2013 στην αρχή της υπόθεσης όπου δεν είχαμε λάβει απάντηση ότι μόνον ε, μία, ε, μόνο ένα αίτημα ε, έγινε αποδεκτό ε, ενός από τους όσους καταδικάστηκαν 9 ετή κάθριξη. Βεβαίω στην Ευρώπη υπάρχει το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη. Είναι μια υπόθεση μεταξύ δικαστών, όπω ξέρετε. Και έτσι έγινε και η σύλληψη τη Ντεσόζα στη Λισαβόνα. Πρέπει να πω πάντως ότι στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιταλίας υπάρχει μια διμερής συμφωνία με, ε, πέραν των πολυμερών που προβλέπει και επιτρέπει την έκδοση πολιτών έχουν εκδοθεί Ιταλοί από την Ιταλία, αλλά δεν μπορώ να πω εδώ ότι υπάρχει ισχυρή πίεση για το θέμα αυτό, αλλά ούτε και συζήτηση πραγματικά για το κατά πόσο είναι παράλογη ή τέτοια πρόβλεψη. Θα μπορούσαμε ίσως να έχουμε εξασφαλίσει και το αντίθετο για τον αριθμό των υποθέσεων η μόνη υπόθεση είναι αυτή που σα ανέφερα. Είναι ε, η μόνη που σε οριστικέ καταδίκε και ο ΙΕ λέει ότι είναι και η μόνη υπόθεση παγκοσμίω. Τώρα, ε, από όσα έχουμε συλλέξει από τον τύπο θα το δείτε και στο έγγραφο που σα έχω στείλει, προσωπικά πηγαίνοντα στην Ισπανία όπου ξεκίνησε ε, από 12 ανακριτέ, όχι από την εισαγγελία η υπόθεση, πήγα στην Ελβετία Πήγα στη Γερμανία για την υπόθεση Ρέιμσταϊν. Ε, στην Ιταλία τέλος πάντων ήταν η μόνη υπόθεση που οδήγησε σε τελική καταδίκη και είναι σαφές η κοινή γνώμη δεν γνωρίζει καλά τα θέματα αυτά. Έχουν γίνει και κάποια απίστευτα σχόλια και από άτομα μέσης ή ανώτερης μόρφωσης. Διάβασα και μία συζήτηση που έγινε εδώ στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Ίσως κάποιος ταλός βουλευτής με αφορμή την έκθεση Φέινσταϊν είχε πει κάτι που κανείς θα ήθελε να... θα περίμενε να έχει καταλάβει κάποια περισσότερα, αλλά τα θεωρώ αδιανόητα αυτά σε δημοκρατικά καθεστώτα. Δεν μπορούμε να παραγνωρίζουμε τη σημασία των ε, ε, υποθέσεων αυτών, διότι αλλιώ θα είμαστε ιονοί δημοκρατίε. Αν θέλουμε να είμαστε πραγματικώ δημοκρατικοί, πρέπει να προχωρήσουμε. Πάντω, αυτά ε, τα γεγονότα, τα φασανιστήρια λόγω χάρη αυτά, όχι απλώ ήταν τελείω περιτά, όπω είπε η έκθεση Πένσταϊν, αλλά δεν μπορούμε και να τα επιτρέπουμε. Και δημιουργούν απλώ αίτια να προσελητήσουν οι τρομοκρατικέ ομάδε πιο αποτελεσματικά και άλλα μέλη. Άρα, ε, α, ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Κυρία Σιν, παρακαλώ. Thank you. I agree with... Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με τις εξαιρετικές παρατηρήσεις του κυρίου Σπατάρο. Απαντώντας στο ερώτημα που μου τέθηκε όσον αφορά την υπόθεση Αλνάσρη κατά Πολωνίας, είναι σωστό ότι η Πολωνία άσκησε έφεση, αλλά απορρίφθηκε η έφεση και η απόφαση έγινε τελεσίδικη το Φεβρουάριο του 2015. Είναι επίσης σωστό ότι πληρώθηκε αποζημίωση από την Πολωνία στον κύριο Αλνασί. ήθελα όμως και πάλι να τονίσω ότι μιλάμε εδώ για τις πιο σημαντικές παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης και του Διεθνούς Δικαίου. Ε, τα βασανιστήρια απαγορεύονται και ξέρουμε ότι η υπέστη η εικονική εκτέλεση Ε, αναγκαζόταν να στέκεται σε πολύ κακές στάσεις, ε, τα χέρια του σχεδόν ε, εξαρθρώθηκαν και στην Ρουμανία η έκθεση της Γερουσίας σε συνδυασμό με τις πληροφορίες ότι ο κύριος Χάμερπερκ. Η έκθεση ευσίας μαζί με τα στοιχεία του κυρίου Χάμερπερκ δείχνει ότι φαίνεται ότι ο κύριος Αλνάσρη υπέστη rectal feeding όπου ε, πρέπει να σκύψει το άτομο και τον ταΐζουν από το έντερο. Και η CIA χρησιμοποιούσε αυτή την μέθοδο για έλεγχο της ε, συμπεριφοράς ε, των φλεξμένων ε, χωρίς μάλιστα να υπάρχει έλεγχος από γιατρό. Η σοβαρότητα των παραβιάσεων αυτών δείχνουν ότι ε, θα πρέπει να γίνει κάτι και ότι δεν αρκεί η πληρωμή αποζημίωσης ε, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι δεν ε, έγινε η απαραίτητη έρευνα και ότι δεν απαιτήθηκε λογοδοσία. Αυτή η διαδικασία είναι που ε, διασφαλίζει να μην ξαναγίνουν τέτοιες πράξεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους δυο σας. Συνάδελφοι, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας εκπονήθηκε μια αξιόπιστη έκθεση για τις έκτακτες παραδόσεις της CIA. Το ψήφισμα του φετινού Φεβρουαρίου μας καλεί να επικαιροποιήσουμε τα στοιχεία τη έρευνα και τη έκθεση, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση τη Ειδική Επιτροπής Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η σημερινή ακρόαση αποτελεί μέρος της, αντα... της ανταπόκρισή μας σε αυτό το αίτημα. Νομίζω ότι ήταν εξαιρετικέ οι παρεμβάσει που ακούσαμε σήμερα και όπως επίσης και οι παρεμβάσεις των Ευρωβουλευτών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διότι είναι πολύ δύσκολο και επίμαχο το θέμα. Χαίρομαι που διαπιστώνω ότι κάνουμε το χρέος μας όσον αφορά τη λογοδοσία και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση το κράτος δικαίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, που το κάνουμε αυτό. Οι συντονιστέ και η Επιτροπή στο σύνολό τη θα εξετάσει τι περαιτέρω δράση θα αναλάβουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω του ομιλητέ που βρέθηκαν εδώ σήμερα και όλου του ενδιαφερόμενου που συμμετείχαν στι εργασίε. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, ε, σα ευχαριστώ όλου. Uh, oh, κύριε Σπατάρο, όχι, μεταδίδεται στο διαδίκτυο. μεταδίδεται στο διαδίκτυο η συνεδρίαση. Λοιπόν, σας άκουσαν σίγουρα οι Ιταλοί όσο μιλούσατε. Μεταδίδεται. Να με συγχωρείτε όσο παρακολουθούσατε. Ακόμη και ο κύριος Φάβο μπορεί να παρακολουθούσε ενώ μιλούσαμε. Βέβαια περισσότερο είναι στον υπολογιστή τους από ότι εδώ, είναι αλήθεια αυτό, αλλά έτσι είναι ο κόσμος μας. Colleagues, if you are going to stay, we're going to... Λοιπόν, συνάδελφοι, να παραμείνετε. Έχουμε και άλλο θέμα. Είναι η Επιτροπή Λίμπε. <laughs> Έχουμε μια πολύτιμη μισή ώρα τώρα και το θέμα υπαριθμών 11 στην ημερησία διάταξη. Έτσι εργαζόμαστε, ξέρετε, ε, στην Επιτροπή μας. Πάμε. Λοιπόν, έχουμε το σημείο 11. Από τις 12 μέχρι το 12.30 θεώρηση ενίου τύπου έχουμε πάρα πολλή δουλειά και πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας και θα πρέπει να προχωρούμε κανονικά έτσι, για τους συναδέλφους που θέλουν να περιμένουν. Βλέπω ότι είναι εδώ παρούσα εισηγήτρια και χαίρομαι πάρα πολύ ε, την Σίλβια Ιβόν Κάουφμαν. Κάτι ορίζω. Έχουμε παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορά την πρόταση τροποποίηση του κανονισμού ε, για τη ε, θεώρηση διαβατηρίων. 20 χρόνια ε, κυκλοφορεί ένα είδος, ένα αυτοκόλλητο ε, Visa Sticker, το οποίο παραποιείται και χρειάζεται νέα στοιχεία για βελτιωμένη ασφάλεια, με νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Θα δώσω το λόγο παρακαλώ τώρα στην κυρία Σίλβια Ιβανά Κάουφμαν. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κλοντ, αγαπητέ Πρόεδρε. Το είπατε. Εδώ και 20 χρόνια έχουμε νέα θεώρηση νέου τύπου ε, αυτοκόλλητο και αυτό είχε ξεκινήσει από τη διακρατική συνεργασία από το Σέγγεν και ε, στη συνέχεια ένα κανονισμό του 1995 όπου όλα τα κράτη-μέλη αλλά και η Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτεστάιν και η Ελβετία που συμμετέχουν στο χώρο Σέγγεν συμφώνησαν να κάνουν ε, ε, μια θεώρηση νέου τύπου. Ο κανονισμός αυτός του 1995 στο μεταξύ έχει αλλάξει δύο φορές, το 2002 συγκεκριμένα αλλά και το 2008 και περί τίνος πρόκειται για υψηλά πρότυπα ασφαλείας, φωτογραφία φερρυπίν, να συμπεριλαμβάνεται η, ε, ε αρρύθμιση και το σύστημα ΣΥΣ, με ναι, ΒΙΣ μάλλον για τις ε, βίζες. Το 1995 ε, ήταν η πρώτη εκδοχή του κανονισμού και παρόλες τις αλλαγές που έγιναν τα τελευταία χρόνια, είναι νέα η πραγματικότητα. Εξού και κάνει πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δυστυχώς υπάρχουν πολλές ε, παραποίησεις και στα πολύ ψηλού επίπεδου σε κάποια κράτη-μέλη, με πλαστές θεωρήσεις λοιπόν και αν δεν είναι ασφαλής η θεώρηση νέου τύπου θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τη βλαστογραφία και την απάτη. Το 2009 λοιπόν συστήθηκε μια υποεπιτροπή για να εκπονήσει ένα νέο σχέδιο έναν τύπου και 6 χρόνια χρειάστηκε για να φτιάξει μια νέα βίζα Τώρα επιτέλους τη σχεδιάσανε με νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας, ενιαίο design και το ίδιο ε, χαρτί. Λοιπόν, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες φυσικά, ε, να αναφερθώ σε μερικά σημεία μόνο. Πρώτον, για ποιο λόγο δεν προτείνεται αναθεώρηση του κανονισμού και πάλι. Διότι όταν αλλάζεις για τρίτη φορά σημαντικά ένα κανονισμό, προτείνεται να ξαναγραφεί από την αρχή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν το θέλει αυτό, διότι σημαντικότερες αλλαγές είναι στην απόφαση, την εκτελεστική, δηλαδή τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές, οπότε δεν τίθεται θέμα αλλαγής του ε, ε, νόμου, του κανονισμού επροκειμένου. Προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν το εξής. Εννιά μήνες μετά την έγκριση του κανονισμού να αποκτήσουν ισχύ τα νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας αλλά επί ένα εξάμεινο να ισχύουν και τα παλιά χαρακτηριστικά της θεώρησης νέου τύπου. Αυτό το χρονοδιάγραμμα νομίζω είναι καλά στοιχειοθετημένο από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από τη μία θα πρέπει να βρούμε γρήγορα και να δράσουμε γρήγορα τώρα για να εξασφαλίσουμε τις θεωρήσεις, ε, για να μην μπορούν να παραποιούνται και να πλαστογραφούνται. Από την άλλη πρέπει να δώσουμε και κάποιο χρόνο στα κρατη για να προετοιμαστούν. Ένα τελευταίο υπάρχει εξή κατάσταση. Φαίνεται δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο κατά πόσο η Μεγάλη Βρετανία, η Ιρλανδία και η Δανία θα θελήσουν να συμμετέχουν. Μέχρι τώρα έχουμε όλα τα κράτη-μέλη, συν τις άλλες χώρες έγκεν που δεν είναι κράτη-μέλη της Ένωσης, που έχουν τη θεώρηση νέου τύπου. Και ελπίζω πάρα πολύ να συνεχίσει αυτό να ισχύει τα τρία κράτη ε, αυτά, η ε, Μεγάλη Βρετανία, η Ιρλανδία και η Δανία να συνεχίσουν να συμμετέχουν. Γιατί δεν γίνεται μετά από τόσο καιρό που έχουμε ενιαίες θεωρήσεις, τώρα να αρχίσει ο καθένας να κάνει τη δική του. Ε, οπότε ελπίζω να συμμετέχουν στο γενικό σύστημα. Επίση θέλω να πω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χρειάζεται επιγόντως να δράσουμε και ελπίζω σε μια διαδικασία ε, γρήγορη για να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ η θεώρηση ενίου τύπου καινούργια. Ευχαριστώ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μην εδώ κάποιος συνάδελφος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την εισηγήτρια. Μου πήρε τα λόγια από τη γλώσσα. ε, ε θα ήθελα να συμπληρώσω κάποιες παρατηρήσεις. Πράγματι, το 2009 στην ε, Επιτροπή του άρθρου 6 της Κομισιόν ε, υποστηρίχθηκε ότι θα πρέπει να σκεφτούμε νέα διαμόρφωση της αυτοκόλλητης θεώρησης. Έχουμε επιταχύνει τις διαδικασίες διότι ε, έχουμε διαπιστώσει ότι πάνω στα κάτι μελη ε, αρκετές πολύ πετυχημένες ε, πλαστογραφίσεις. Όπως λοιπόν είπε η συγγήτρια, στην πρόταση έχουμε υιοθετήσει σχετικά σύντομη προθεσμία υιοθέτησης κάποιες τεχνικές παρατηρήσεις στην πρότασή μας. Βλέπετε ότι προβλέπονται δύο νέα μέτρα. Εάν τα κράτη-μέλη συμφωνήσουν ότι είναι απαραίτητο, ε, να έχουμε barcode και αυτό δεν αποτελεί μέρος της παρούσας πρότασης, αλλά δίδεται η δυνατότητα σε μελλοντική ε, απόφαση να έχουμε ένα ε, barcode 2D και και άλλες δυνατότητες εφόσον διαπιστώσουμε πάλι μεγάλο αριθμό ε, πλαστογραφήσεων. Ίσως θα έπρεπε να κάνω μια σύντομη παρατήρηση σχετικά με το γιατί. Προτείνουμε πάλι η αυτοκάλυπτη θεώρηση να είναι σε χαρτί. Εφόσον έχουμε το σύστημα πληροφόρησης για τις θεωρήσεις και το οποίο θα είναι διαθέσιμο σύντομα σε όλες τις χώρες του κόσμου. Όπως πιθανότατα γνωρίζετε, οι θεωρήσεις τύπου D που περιορίζονται στο έδαφος του ενός κράτους μέλους δεν εισάγονται στο σύστημα πληροφόρησης για τις θεωρήσεις. Πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς να καταργήσουμε την θεώρηση σε χαρτί. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να προτείνουμε τροποποίηση του αυτοκόλλητου. αν σε κάποια χρόνια διαπιστώσουμε την καλή λειτουργία του συστήματος πληροφόρησης για τις θεωρήσεις, θα μπορέσουμε να ξανασκεφτούμε. Μήπως θέλουμε να έχουμε μόνο ηλεκτρονικές θεωρήσεις. Κατά τη γνώμη της Κομισιόν όμως είναι πολύ νωρίς ακόμα για κάτι τέτοιο. Νομίζω μπορώ να κλείσω εδώ. Είμαι στη διάθεσή σας αν έχετε ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Thank you very much. We have one... Ευχαριστώ πολύ. Ένα σκιώδη έχουμε, είναι και ο Σαβάρμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την εισηγήτρια. Δεν έχω να πω τίποτα δραματικό. Απλώς ε, μιλώ για να ε, ανταποκριθώ στο καθήκον μου ως και ο να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το έργο της, το μέχρι τώρα, το είναι και το επόμενο. Ε, θέλω να αναφέρω λίγα πράγματα μόνο. Συμφωνώ ότι επήγει το θέμα και χρειάζεται ταχύτατη διαδικασία ακριβώς επειδή είχαμε τόσες πολλές πλαστές ε, θεωρήσεις και μάλιστα πάρα πολύ υψηλού τεχνολογικού επίπεδου, πάρα πολύ άρτιες. Για τον ίδιο λόγο συμφωνώ και με την επιχειρηματολογία αυτή. Να αποκλίνουμε από τον στάνταρ κανόνα, να υπάρξει αναδιατύπωση του κανονισμού. Δεν χρειάζεται τώρα να ξαγραφτεί ο κανονισμός από την αρχή. Συμφωνώ και με τα κίνητρα και με τα επιχειρήματα που δόθηκαν. Υπάρχει και ένα θέμα, δεν είναι, είναι ουδέτερος προς τον προπολογισμό, δεν είναι, οικονομικό το ζήτημα, οπότε μπορεί να ακολουθηθεί η ταχεία διαδικασία και στο Κοινοβούλιο. και καλό είναι να έχουμε και μια προθεσμία εξάμεινη ε, για την αντικατάσταση. Τίποτα άλλο να ε, προσθέσω. Η Σίλβια Ιβών, συγγήτρια. Όχι. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι ε, ειλικρινά την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γιατί πρέπει να υπάρχει χαρτί αυτό το αυτοκόλλητο είναι πάρα πολύ σημαντικό επιχείρημα να το λάβουμε υπόψη μας και πολύ καλό ε, το γεγονό ότι έχει ε, προβλέψει και προνοήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν χρειαστούν επιπλέον νέα τεχνικά χαρακτηριστικά να μπορούν να συμπεριλαμβάνονται όλα αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Να προχωρήσουμε γρήγορα όμως, γιατί το θέμα ε, πήγε. Ευχαριστώ πολύ Σίλβια Ιβών και σε ευχαριστώ που παραμείνες στο τέλος της ακρόασης για να μπορέσουμε να δούμε το θέμα σου σήμερα το πρωί. Ευχαριστώ. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά για να προχωρήσει η μερίσια διάταξη. Λοιπόν, σας είπα και το πρωί και επαναλαμβάνω ότι η συνεδρίασή μας το απόγευμα θα αρχίσει στις 3.30 δηλαδή για τις 3 και οι ψηφοφορίες αναβάλλονται. Ένα mail έχει σταλεί σε όλα σας τα γραφεία. Ευχαριστώ πολύ.